Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητοί κυρίε και κύριοι, σα καλωσορίζω θερμά στη συνεδρίασή μα τη ε, εβδομάδα αυτή από την Βρέμη και την Νότια Σαξονία έχουμε ένα, την κάτω Σαξονία, συγγνώμη, ένα γκρουπ επισκεπτών είναι επισκέπτες της κυρίας Κεζίνε Μάης. Ναι, καλώς ορίσατε. Μπορεί να εγκριθεί λοιπόν η μερίσια διάταξη, αν δεν έχει κανείς καμία αντίρρηση ή ένσταση. Και τα ε, πρακτικά επίσης, της 31ης 8 2015, εάν δεν διαφωνεί κανείς σας. Ερχόμαστε λοιπόν στην έκθεση για τα drones, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είναι η συγγήτρια κυρία Τζακλίν Φώστερ και αύριο η ψηφοφορία θα δώσουμε αμέσως το λόγο στην συγγήτρια. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαστε σε θέση να ε, συζητήσουμε πλέον αυτό το θέμα για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Θα ψηφίσουμε αύριο. Είναι ε, πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε να παραμείνουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δουλέψουμε στο πλαίσιο του πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αεροπορία καλό είναι να μην καθυστερήσουμε, να ε, περάσει στην Ολομέλεια τη δεύτερη του Οκτωβρίου. Βέβαια πρέπει πρώτα να περάσει το θέμα από την δική μας Επιτροπή και δεν θεωρώ ότι αυτό είναι δεδομένο. Είμαι ε, σίγουρη ότι οι περισσότεροι ε, εξημών θα ε, είστε και στο Στρασβούργο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά τις, ε, την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε κατά τους τελευταίους μήνες. Θα ήθελα απλώς να πω ότι η ουσία βρίσκεται στον τίτλο και είναι για ασφαλή χρήση. Μιλάμε λοιπόν για την ασφάλεια, την ασφαλή χρήση των RPAs ε, των συστημάτων ε, τηλεκατευθυνωμένων αεροσκαφών, των μη επανδρομένων ε, αεροσκαφών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Συμπεριλαμβάνει τα πάντα από την κατασκευή μέχρι την αλυσίδα ανεφοδιασμού και εμείς έπρεπε να δούμε πώς λειτουργεί κάτι τέτοιο, πώς μπορούμε να ε, δούμε την ανάπτυξη των χρήσεων των drones, των μη επανδρομένων αεροσκαφών και μιλάω για μη στρατιωτική χρήση, δεν μιλάω για τη στρατιωτική χρήση, αυτό το τονίζω, πρόκειται για την μη στρατιωτική χρήση και περί αυτού ακριβώς ε, πρόκειται, ε, γι' αυτό ακριβώς, αυτό πραγματεύεται η δική μας γνωμοδότηση. Ένα πλαίσιο ιδεών μεταφορών. Εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών θέλουμε ε, οι ρυθμιστές, η Επιτροπή, ε, όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτό το θέμα και οι εθνικές κυβερνήσεις βεβαίως, ε, τα Υπουργεία Μεταφορών, τα τμήματα ασφαλείας κλπ. Όλα αυτά ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, στη συγκεκριμένη έκθεση και γι' αυτό ακριβώς ε, τα έχουμε συμπεριλάβει. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθεριών κατέθεσε μία γνωμοδότηση. Εγώ μίλησα με την... Με η κυρία Ντάνχαν, η οποία η υπέβαλε την γνωμοδότησή της, αλλά μίλησα με εκείνη πριν γίνουν οι, τροποθε, τροπολογίες, πριν από την εβδομάδα του, ε, της Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Μετά έπρεπε βέβαια να περιμένουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε εδώ σήμερα. Οπότε ε, ό,τι έχει εκφράσει ως άποψη η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει συμπεριληφθεί ε, στη συγκεκριμένη έκθεση. Και θα ήθελα να πω ως προς τη δική μου προσέγγιση είναι πραγματικά μία ε, άποψη η οποία προσπάθησε να συγκεράσει τις απόψεις όλων των πολιτικών ομάδων. Δεν είναι πολιτική χαρακτήρα η έκθεση. Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουμε οι σκιώδεις εισηχητές όλων των πολιτικών ομάδων ήταν εξαιρετικοί, ήταν επικοδομητικοί. 153 τροπολογίες ε, τις οποίες ε, χτενίσαμε ε, και καταλήξαμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Ο τρόπος με τον οποίο καταλήξαμε στις συμβιβαστικές τροπολογίες ήταν πάρα πολύ όριμος υπήρξαν ορισμένα πράγματα τα οποία θα ήθελα εγώ να είχαν ε, επιτευχθεί αλλά δεν τα ε, κατάφερα. Κάποιοι ήθελαν ορισμένα πράγματα να ε, διαγραφούν, δεν τα κατάφεραν. Υπήρξε ένα πνεύμα συμβιβασμού. Είναι πάρα πολλές οι τεχνικές λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά το το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν του σκιώδει εισηγητέ αλλά και του συναδέλφου από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, οι οποίοι ήταν και εκείνοι πάρα πολύ επικοδομητικοί. Δεν θα ήθελα να πω πολύ περισσότερα, αλλά σε τομεί ε, που αφορούν για παράδειγμα τους, ε, τις, τις, τον τομέα τον κατασκευαστικό των drones. Ε, εμείς ε, έχουμε επιχειρήσεις πολύ μεγάλων συμφερόντων. Θέλουμε βεβαίως να μπορούμε να πολλούμε τα προϊόντα μας στα, στον υπόλοιπο κόσμο. Θέλουμε βεβαίως να υπάρχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να το πούμε και αυτό. Είμαστε και πολύ μεγάλη αγορά. Πώ θα το κάνουμε όμω αυτό, δεν θα μπω σε πολλέ λεπτομέρειε. Όμω πρέπει να βασιστούμε σε αυτό που οι Εθνικέ Υπηρεσίε Πολιτική Αεροπορία προσπαθούν να κάνουν, ε, ε, να μην ξεχνάμε τον Τζάρου, να μην ξεχνάμε την ΕΑΖΑ που είναι Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλεια Αεροπορίας. Η ΕΑΖΑ ε, συμμετέχει στον Γιάρου. Είναι λοιπόν αυτό πάρα πολύ σημαντικό και όλο αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε ε, με έναν απλό τρόπο για τα θέματα της προστασίας των δεδομένων, της προστασίας του ιδιωτικού βίου. Θέλουμε να είναι πολύ ισχυρό το κείμενό μας ως προς αυτό, να αισθάνεται εμπιστοσύνη το κοινό ότι δεν υπάρχει ε, πρόβλημα με την προστασία των δεδομένων, να μην φοβάται ο κόσμος και όταν βλέπουμε ας πούμε τη λειτουργία των μη επανδρομένων αεροσκαφών υπάρχουν ε, έμποροι ε, οι οποίοι έχουν ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο, είναι πάρα πολύ ικανοί, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό το θέμα. Ξέρουμε όμως ότι σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν και ανόητοι, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πολύ διασκεδαστικό να παίζουν με τα drones και βεβαίως πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει καταχώρησή τους, ότι υπάρχει αδειοδότηση, ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις εκπαίδευσης ε, όσων ε, τα ε, χρησιμοποιούν οπουδήποτε. Εντάξει, βέβαια μιλάμε για έναν ε, γεωργό σε κάποια γεωργική ε, εκμετάλλευση, είναι κάτι διαφορετικό. Ε, θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια συνολική προσέγγιση, δεν θέλουμε να δέσουμε και χειροπόδαρα τους ρυθμιστές και να τους βγάλουμε σε μια θέση στους οποίους χωρίς να γνωρίζουν τι, μπορούν χωρίς να γνωρίζουν τι είναι αυτό που θέλουμε και να τους εμποδίσουμε να προβούν στις τεχνολογικές ε, ε, εξελίξεις ε, στις οποίες πρέπει να προβούν. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση που θα είναι επικερδής για όλους. Αυτά λοιπόν από μένα. Φαντάζομαι ότι οι σκιώδεις εισηγητέ θα έχουν και εκείνη σχόλια. Χαίρομαι που εκπροσωπείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Τζάκι Φώστερ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γνώμη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά την κυρία Φώστερ για το έργο της και τις συμβαστικές προτάσεις που επιτάχυναν στο τέλος τη σύγκληση απόψεων για να υπάρξει συμφωνία σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Δεν θέλω να προσθέσω πολλά στα όσα είπε η ίδια, να την ευχαριστήσω και τώρα θα πρέπει γρήγορα να τελειώνουμε αυτή η ιστορία, να την ολοκληρώσουμε. Συμφωνώ με όλα όσα είπε για το πλαίσιο, αλλά το πλαίσιο είναι ένα λευκό χαρτί και είναι για όλους μας πολύ δύσκολη η διαδικασία και μπορεί να είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητέ, αλλά θα πρέπει να το ε, γράψουμε αυτό το πλαίσιο, να το δημιουργήσουμε, γιατί δεν υπάρχει ακόμα. Και υπάρχει και τεράστια ηλικιώδης ε, ταχύτητα, αχαλήνωτη φαντασία ε, των δημιουργών και άπειρες εφαρμογές παντού, στην εστίαση, στο delivery, στην ψυχαγωγία, στη διασκέδαση. Είναι όνο και αριθμό, οι εφαρμογέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ε, προηγηθούμε. Χαίρομαι τώρα επί της ουσίας για το ευρωπαϊκό πλαίσιο, επαναλαμβάνω, αυτό το λευκό χαρτί που θα πρέπει να γίνει μια πρόταση και να την προωθήσουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για μένα γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στην ε, ψυχαγωγική και στην επαγγελματική χρήση ε, των ε, μη επανδρομένων αεροσκαφών. Θα πρέπει να ε, υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο κανόνων και να προσαρμόζει την νομοθεσία ανάλογα με τον κίνδυνο που συνιστά κάθε δραστηριότητα. Παράδειγμα, στους αυτοκινητοδρόμους και τα ΙΟΤΑΧΗ ε, και τα φορτηγά έχουν τον ίδιο κώδικα δικής κυκλοφορίας αλλά χρειάζονται διαφορετική άδεια και άδεια οδήγησης. Επίσης, ε, Υπάρχουν και ε, πολιτικά τέτοια αεροσκάφη. Ο κόσμος όταν ακούει drones νομίζει ότι είναι στρατιωτικά και θεωρεί ότι είναι κατασκοπία. Δεν θα πρέπει να το φοβούνται. Ίσως να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα που μπορεί να σας φανεί παρατραβηγμένο. Όταν εφευρέθηκε ε, η φωτογραφική μηχανή, υπήρχε και το zoom. Αλλά δεν σημαίνει ότι πήγαινε και τραβούσε φωτογραφία το γείτονά σου στη βυσίνα του. Ε, η προστασία λοιπόν των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής είναι δεδομένη και ε, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος κάνει τι κάθε φορά. Θα πρέπει λοιπόν να ε, προστατεύσουμε και τις ε, πτήσεις ε, που είναι εκτός οπτικού πεδίου. Είναι μόνο τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη που κάθε φορά ο χειριστής τα βλέπει. Ε, σας λέω είναι τρομακτικές οι εξελίξεις στην τεχνολογία, πρέπει να το προβλέψουμε. αν θέλουμε όμως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ΕΑΣΑ να έχει λόγο για κάθε είδους ε, τηλεχειριζόμενα ή τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη θα πρέπει να έχει και τους απαραίτητους εκείνους πόρους. Να μην έχουμε γραφειοκρατικά εμπόδια ε, με εχώριση μεν αρμοδιοτήτων σε μια ανώτερη αρχή που δεν θα έχει όμως τις δυνατότητες να εκτελέσει την αποστολή της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και για τις θέσει εργασίας και για τη δημιουργία τέτοιων θέσεων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, κύριος Γιάννης Σέμκε. Ε, Θα ήθελα, ξεκινώντας να πω το εξής, ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το θέμα αυτό συζητιέται για πρώτη φορά. Και αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η έκθεση αυτή να είναι ποιοτική. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που μετά από εβδομάδες αλλά και μήνες ολόκληρους, ε, επιτέλους καταλήξαμε σε μια καλή έκθεση. Σέβομαι ιδιαίτερα τη δουλειά της ε, κυρίας ε, Φώστερ, η οποία τελικά προέκυψε από πάρα πολλές τροπολογίες. Αρχικά είχαμε 153 τροπολογίες, 20 είχαμε από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και τώρα λοιπόν έχουμε 30 συμβιβαστικές ε, προτάσεις και θέλω να προτείνω στους συναδέλφους από τη Σοσιαλιστική Ομάδα να στηρίξουν αυτές τις ε, προτάσεις. Στη συνάντησή μας ε, το βράδυ σήμερα θα το προτείνω αυτό στην πολιτική ομάδα. Νομίζω λοιπόν ότι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη όχι μόνο εξελίσσονται ταχύτατα ως τεχνολογία, αλλά εγκυμονούν και ένα κίνδυνο, διότι αυτή η νέα τεχνολογία συνεπάγεται και κινδύνους. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε αυτούς τους κινδύνους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια. Κάθε ημέρα ακούμε στις ειδήσει ότι κοντά ε, στα αεροδρόμια εμφανίζονται κάποια μη επανδρομένα αεροσκάφη και αρχίζουμε να τρέμουμε γιατί φοβόμαστε μην υπάρξει κάποια σύγκρουση. Και καταλαβαίνετε ποιες θα είναι οι συνέπειες ε, αυτού του ενδεχόμενου της σύγκρουσης. Και υπάρχει και ένας δεύτερος κίνδυνος. Πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ε, χρησιμοποιούνται εκμεταλλεύονται ε, διάφορες εταιρείες ε, για να συγκεντρώσουν στοιχεία για την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Αυτό προφανώς απαγορεύεται από τον νόμο. Και υπάρχει και άλλο ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και συγκεκριμένα το κατά πόσον οι κανονισμοί της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να αφορούν μόνο στην εμπορική χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών ή κατά πόσον θα πρέπει να αφορούν ε, και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται ως χόμπι κατά διάρκεια του ελεύθερου χρόνου ψυχής και το καθεξής. Στην πρώτη περίπτωση δεν πρέπει να είμαστε Μάλλον σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη ενοχή. Είναι διάφορο το γιατί χρησιμοποιείται ένα τέτοιο μη παντρωμένο σκάφο. Γιατί για όποιο σκοπό και αν χρησιμοποιείται, αν συγκρουστεί με ένα κανονικό αεροσκάφο, καταλαβαίνετε οι συνέπειε παραμένουν οι ίδιε. Όσον λοιπόν ε, αφορά σε αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του μοντελισμού ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και τέλος επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που σύντομα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες μας και έχω και μία παράκληση προς τον ε, κύριο Πρόεδρο ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πει ε, τι ακριβώς έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Αυτά που έχουμε προετοιμάσει εμείς είναι πάρα πολύ καλά, αλλά οι νομικές προτάσεις ε, κατατίθενται από την Επιτροπή. Πάρα πολύ ωραία. Προφανώς και τελειώνει η συζήτηση. Η Κομισιόν έχει πάντα το λόγο ε, η οποία μπορεί και να μιλήσει ελεύθερα και ελπίζω να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα θέματα. Ο κύριος Ματέη Φων Μίλτεμπεργκ ε, από του φιλελευθέρου, Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Φώστερ για την εξαιρετική τη εργασία αλλά και του υπολείπου και ηγητές για ε, ε, την συνεργασία. Ήταν πολύ στενό το χρονοδιάγραμμα και έπρεπε να έχουμε πάρα πολύ σαφείς συμβαστικές τροπολογίες αλλά νομίζω ότι κάναμε καλά τη δουλειά μας. ελπίζω και βοήθησε η κυρία Φώστερ ότι στην αγγλική βιβλιογραφία στο μέλλον θα υπάρχει μια πολύ γνωστή φράση, περίφημη και όχι το να ζει κανείς ή να μην ζει, αλλά το να έχει κανείς ντρόν ή όχι ντρόν και να τα χρησιμοποιεί και με ποια ε, πλαίσια και ποιους όρους και προϋποθέσεις. To drone or not to drone λοιπόν. Η απάντηση είναι καταφατική ε, και ε, ε, μας ενδιαφέρει το πλαίσιο που θα τεθεί στην ΕΑΣΑ για τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τις πτήσεις αυτών των αεροσκαφών στην Ευρώπη. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΛΥΒΕ που τονίζει τη σημασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων. Είναι πάρα πολύ καλή κατά την άποψή μου η γνωμοδότηση αυτή και μια που συζητούμε για τις τροπολογίες εγώ θα ήθελα να υιοθετήσουμε την ε, γνωμοδότηση της ΛΥΒΕ, έτσι και αλλιώς στις συμβαστικές τροπολογίες πολλά έχουν ήδη ενσωματωθεί. Μια που μιλάμε και για συμβαστικές τροπολογίες, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάντα συμβιβασμός και καμιά φορά χρειάζεται μετά από έλεγχο ή μετά από ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο να επέλθουν κάποιες διευκρινήσεις. Αύριο θα κάνω τροπολογίε προφορικές, σας το λέω από τώρα για να μην εκπλαγείτε, ε, στη συμβαστική υπαριθμών 9 ας πούμε και αφορά την παράγραφο 20 θα ήθελα να εκφράσουμε την εξή θέση. Όταν μιλούμε για ε, drones ε, που πετούν εκτός οπτικής επαφής θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, ανείχνευσης και ε, παράκαμψης. Ε, ε, με τεχνολογία δηλαδή να μπορεί κανείς να, τα ε, καταγράφει και να τα παρακάμπτει όταν δεν τα βλέπει αυτά τα αεροσκάφη. Και υπάρχουν και τροπολογίες για την εφαρμογή των κανονισμών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν συζητούμε για νομοθεσία και κανονισμούς τουλάχιστον αν μη τι άλλο, να καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αρχίσουν τουλάχιστον να προβληματίζονται για να βρούμε έναν τρόπο να ενισχυθεί η μελλοντική νομοθεσία. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξή σας αγαπητά μέλη της Επιτροπής μας και για την τροπολογία 133 καθώς και την 134 που αφορούν αυτά τα θέματα της εφαρμογής μελλοντικής νομοθεσίας για τα drones. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κίλονεν. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ. Η Κατορίνα Κονέτ ε, είναι, ήταν σκιώδης εισηγητής. Ε, θα σας διαβάσω τα εξής. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος ε, που καταλήξαμε σε καλές συμβιβαστικές τροπολογίες και επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε αύριο με την ψηφοφορία. Ε, θα γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το θέμα των drones δεν το θεωρούμε μόνο ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά ως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα όταν πρόκειται για την παρακολούθηση και την κατασκοπία. Πρέπει να γνωρίζει η Επιτροπή ότι η τεχνολογία οποία ε, εξελίσσεται τόσο ραγδαία που είναι αδύνατον για την νομοθεσία να αντιδράσει με αποτελεσματικό τρόπο. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση γιατί τα μία πανδρομένα αεροσκάφη δεν γνωρίζουν σύνορα. Επίσης η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει ε, την ε, εθνική νομοθεσία, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός τρόπος αντιμετώπισης των drones. Είναι τόσο μικρές οι κάμερες σήμερα που μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα υπτάμενο αντικείμενο και αυτό καθιστά την κατάσταση πολύ πιο περίπλοκη. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ τη χρήση των drones για σκοπούς αναψυχής και ε, την ε, ε, μη στρατιωτική χρήση όταν τα drones χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για την αξιολόγηση της, των επιδόσεων στην εργασία. Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζεται το μέσο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πιθανότητα ατυχημάτων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν τροπολογίες που αναφέρονται σε ε, τεχνολογίες ανείχνευσης και αποφυγής, όπως και τη δυνατότητα αναγνώρισης των drones. Αν κάθε ε, κράτος έχει το δικό του σύστημα, αυτό ε, θα ε, δημιουργούσε, ε, δεν θα δημιουργούσε υποχρεωτικά ένα καλύτερο περιβάλλον ασφάλειας για όλους. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη όλες αυτές τις συστάσεις ε, και κυρίως τις συστάσεις της εισηγήτριας της κυρίας Φώστερ. Αυτά εκ μέρους της Καταρίνα. Merci, Monsieur le Président. Η κυρία Καρυμαντελή, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του συναδέλφου του κυρίου Κρέλη Ντέβορ που κολλείεται και απουσιάζει, αλλά ε, τον εκπροσωπώ εγώ εξ ονόματος των Πρασίνων. Ε, κυρία Φώστα, σας ευχαριστούμε πολύ για το έργο σας. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και οι οικολόγοι συμφωνούν με κάποιες συμβαστικές τροπολογίες για θέματα κομβικά για μας και βασικά. Θυμήσατε και θα πρέπει να τονίσουμε κι εμείς ότι Σήμερα χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αυτή όμως η νομοθεσία δεν θα πρέπει να θέτει αναμφιβόλων την προστασία των δεδομένων. Το λέτε και στις τροπολογίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, τα προσωπικά δεδομένα. Εμείς κάναμε μια τροπολογία που την έχετε συμπεριλάβει στις συμβαστικές και έχει ιδιαίτερη σημασία. Και είναι όλα αυτά τα θέματα ε, που έχουν να κάνουν με τις υπερπτήσεις drones σε χώρους και τόπους που θεωρούνται επικίνδυνοι ε, οι στόχοι ε, που είναι εργοστάσια πυρηνικά ή χημικά και τα λοιπά, αυτά τα έχετε συμπεριλάβει στις τροπολογίες σας. Αύριο θα κάνουμε και εμείς μια προφορική τροπολογία για να σας δείξουμε σε ποιο βαθμό αυτή η νέα τεχνολογία μπορεί να είναι χρήσιμη. Έχουμε μια παγκόσμια αναταραχή τώρα ε, ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και drones για να μετρούν την ατμοσφαιρική ρήπανση, για το θόρυβο. Είναι μια προφορική τροπολογία λοιπόν των πρασίνων που θα έρθει αύριο στην ψηφοφορία. Γενικά συμφωνούμε και είμαστε ικανοποιημένοι και βεβαίως θα υποστηρίξουμε όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κριστίν Γοβονταλόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω κυρία Φώστε για την εργασία όλη αυτή που έγινε σε αυτή την έκθεση. Είναι ένα μείζον ζήτημα και πρόκληση για το μέλλον της πολιτικής αεροπορίας. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά και όλους τους κοιόδης αλλά και τους υπολείπους βουλευτές που συμμετείχαν στην εργασία αυτή και για τις συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες βελτιώνουν ουσιαστικά το κείμενο το αρχικό της έκθεσης δείχνουν πόσο ενδιαφέρει αυτό το θέμα όλα τα μέλη της Επιτροπής. Τα ζητήματα ασφαλείας βεβαίως ε, κυριαρχούν και χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση και τον έλεγχο των drones. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω να γίνεται μία διάκριση ανάμεσα ε, ε, στην εμπορική και στην προσωπική χρήση για ψυχαγωγία. Ε, ε, εσωτερική αγορά σημαίνει μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη και για δημιουργία θέσεων εργασίας με πάρα πολύ υψηλή δίκευση. Ε, χρειάζεται ένα πλαίσιο για να υπάρξουν εφαρμογές και χρήσεις σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Είναι καλή αυτή η ευρωπαϊκή επικράτεια ως κλίμακα για να πλαισιωθεί ε, με κανόνες ε, αυτό ο χώρος και με νέους κανόνες για την προστασία των προσώπων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όλα αυτά πολύ ωραία τα έχει υιοθετήσει η έκθεση. Με την έκθεση αυτή έχουμε και την ευκαιρία να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τη βολιδοσκοπήσουμε ως προς τις προθέσεις της. Προσανατολίζεται σε μια ειδική οδηγία για τα drones, σε αναθεώρηση κανονισμού ή σε ένα γενικότερο κείμενο για την ΕΑΣΑ και τις νέες αρμοδιότητες. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα πρέπει να είναι τμήμα του πακέτου για τις αεροπορικές μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δομινίκ Ρίκε. Ευχαριστώ πολύ θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ πως και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι ε, την ε, κυρία Φώστερ που φαίνεται πραγματικά φαίνεται να ε, την χάνει η έκθεση αυτή ευρείας συνένεσης, ομοφωνίας. Είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε δεδομένου ότι έπρεπε να υπάρξει μία ρύθμιση λόγω των θετικών και αρνητικών συνεπειών αυτής της τεχνολογίας και δεδομένου του γεγονότος ότι βέβαια πρέπει να υπάρχει μια ρυθμιση λογω των θετικων και αρνητικων συνεπειων αυτή τη τεχνολογία και προσέγγιση στο τι ακριβώς συνιστά ένα μη επανδρομένος αεροσκάφος. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και για τον έλεγχο των χρήσεων αλλά και για την ενίσχυση ε, της έρευνας και της ανάπτυξης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να έχουμε ένα αρμονισμένο πλαίσιο το οποίο και οι σκιώδεις και η κυρία Φώστερ κατάφεραν να επιτύχουν, αλλά η τεχνολογική πρόοδος είναι καθημερινή σχεδόν, ε, δεν αλλάζει όμως ε, άρδιν τη φύση των προβλημάτων που τίθενται. Οι συνάδελφοι, οι σοσιαλιστές έθεσαν το θέμα αυτό της ασφάλειας ε, μεταξύ άλλων γιατί βρισκόμαστε σε αβέβαιους καιρούς και το θέμα της ασφάλειας μπορεί να ε, θεωρηθεί αρκετά ε, περίπλοκο. Η ικανότητα λοιπόν ανάπτυξης κινητήρων όλο και περισσότερο, όλο και καλύτερων ε, για τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη αυτό μπορεί να έχει ε, αποτέλεσμα αυτό που είδαμε για παράδειγμα στο YouTube ότι ιδιώτες ε, μπήκαν σε τέτοιου είδους αεροσκάφη και έκαναν καταπληκτικές επιδείξεις αυτό βέβαια έχει και αρνητικά το δεύτερο πρόβλημα είναι η διαφορά ανάμεσα στην εμπορική χρήση και την χρήση αναψυχής αν πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα υπάρχει μία επιστροφή των drones ε, ε, που έχουν ξεφύγει από το οπτικό πεδίο απλώς από ένα iPhone, αυτό πραγματικά είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναψηφής. Η πρόοδος λοιπόν που γίνεται όλο και, όλο και περισσότερο στην τηλεκατεύθυνση ε, και σε άλλους τομείς αλλάζουν τη φύση των προβλημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς ισχύει αυτό που είπε η κυρία Φώστερ, ότι πρέπει να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να είναι γενικό, όχι πολύ δεσμευτικό, ε, και το οποίο θα ισχύει ε, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών, ε, της τεχνολογικής προόδου. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα καθήκον, ένα καθήκον και να ε, ε, βοηθήσουμε με το ρυθμιστικό μας πλαίσιο την πρόοδο, ε, αλλά πρέπει και να την πλαισιώσουμε κάπως και νομίζω ότι αυτό το κατάφερε πολύ καλά η κυρία Φώστερη και ελπίζω μόνο καλές εκπλήξεις και όχι τόσες κακές να έχουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Danke sehr. Die nächste ist Marie. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη η Μαρή Κριστίν Νοτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ για την έκθεσή σας που βεβαίως είναι άκρος ενδιαφέρουσα όσο και σημαντική, ιδιαίτερα στο δεδομένο πλαίσιο. Έχω όμως μερικά σχόλια να κάνω. Γιατί ε, νομίζω μπαίνετε στα χωράφια των κρατών μελών εδώ κυρία Φώστερ. Γιατί υπάρχουν στρατηγικά ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση των ντρόουν, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό τομέα και στον αστυνομικό. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την νομιμοποίηση για να επιβάλλει κοινή νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Είπατε ότι καμιά φορά ε, αυτό είναι μεγάλη απειλή για την ασφάλεια των πολιτών, την εδαφική ακαιρεότητα και την εθνική άμυνα, την οποία αγγιάται το κράτος. Γι' αυτό ακριβώς τα κράτη θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να πλαισιώσουν τη χρήση των drones στο έδαφος τους, χωρίς να προσκρούν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, σε αυτή την κατεύθυνση παρακαλώ να καταλάβετε ε, ε την, ε, τις δικές μας τροπολογίες 1381 ε, και 93. Ε, έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που θέλουμε μεν να υπάρχει, αλλά τα κράτη-μέλη να έχουν την ε, πλήρη αρμοδιότητα και ελευθερία για τα drones. Στη συνέχεια, όταν λέμε ότι τα μη επαδρομένα αεροσκάφη μπορούν ενδεχομένω να είναι σοβαρή απειλή, βασίζομαι σε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Α πούμε, πρόσφατα είχαμε υπερπτήσει πάνω από γαλλικά πυρηνικά εργοστάσια που βλέπετε πόσο επικίνδυνο είναι και τη μελλοντική τους χρήση για τρομοκρατικούς σκοπούς που δεν μπορεί βεβαίως να αποκλειστεί. Τονίσατε κυρία Φώστερ τη χρήση των δρόμων στο Ισραήλ, στην παράγραφο 3 το λέτε αυτό και προς την πρόταση ψηφίσματος ακριβώς ε, φαίνεται αυτό που λέω. Ξέρετε ότι ο Ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί αγρίως τα drones, ιδιαίτερα κατά του άμαχου πληθυσμού και σύμφωνα ε, με ε, μία ε, μη κυβερνητική οργάνωση για τα παιδιά στην Παλαιστίνη, 164 παιδιά έχασαν τη ζωή τους από τέτοιες επιθέσεις το 2014 στον πόλεμο στη Γάζα. Και είμαστε και βέβαιοι ότι κάνουν και υπερπτήσεις από το Ισραήλ ο στρατός στη Συρία χωρίς την παραμικρή άδεια και έγκριση. Για να καταλάβετε πόσο στρατηγικό είναι αυτό, παρακαλώ αυτό το παράδειγμα για το Ισραήλ αναπτύσσεται στην παράγραφο 3 και ε, υπό την έννοια αυτή θέσαμε και εμείς την τροπολογία υπαριθμό 42. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πέτερ Λούντ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ε, και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ την κυρία Φώστερ για την πολύ καλή δουλειά. Η διαφορά ανάμεσα στον ελεύθερο χρόνο και στην επαγγελματική χρήση και τις διάφορες δυνατότητες ελέγχου οποτεδήποτε τα μη επανδρομένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για μη επαγγελματικού ε, σκοπούς. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια αγορά η οποία τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει τεράστια αύξηση. Έχουμε το μοντελισμό, τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για ε, τέτοιου είδου δραστηριότητε ή και άλλα μη παντρωμένα σκάφη που χρησιμοποιούνται για να γυρίσουν φιλμ για να βγάλουν φωτογραφίε. Έχουμε αεροσκάφη ε, τα οποία ε, αγοράζονται για ιδιωτικούς σκοπούς, όπως σας είπα, για να βγάζουν φωτογραφίες ή να γυρίζουν φιλμ. Όλα αυτά είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Και βεβαίως ε, είναι και το θέμα της ιδιωτικής ζωής. Γιατί όταν ένα τέτοιο μη υπανδρομένο αεροσκάφος πετάει πάνω από τις ε, ακτές, πάνω από τις ε, πλάζ, πώς μπορεί κανείς να ελέγχει αυτά τα αεροσκάφη. Τα μη υπανδρομένα αεροσκάφη έχουν την τεχνολογία με την οποία είναι εξοπλισμένα Υπάρχουν όμως ε, και την αντίγραφα. Τα επίσημα είναι πάρα πολύ ακριβά και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορεί κανείς να ελέγξει ε, το ότι θα υπάρχει κοινωνική νομοθεσία που θα ελέγχει τα πάντα. Και τα αεροδρόμια θα μπορούσαν να περιοριστούν μόνο για τις πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας, αλλά αυτό είναι λιγάκι δύσκολο. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Τζάκη Φώστερ και όλους όσοι έλαβαν μέχρι τώρα το λόγο. Εγώ θα ήθελα να συνέχισε και που σταμάτησε η κυρία Ρικέ, ότι πράγματι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια νέα εξέλιξη η οποία χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς, ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κατασκοπία και ε, ιδιωτική και στρατιωτική. Αυτό μπορεί να απαγορευτεί με τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων. Όμως μπορεί κανείς και να τα χρησιμοποιεί επαγγελματικά για πράγματα που ακόμα δεν υπάρχουν. Ας πούμε, μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει για έλεγχο κυκλοφορίας ή μπορεί να τα χρησιμοποιεί και για παιχνίδι ε, το είπε αυτό και η κυρία Φώστερ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο για καινοτομία και στην Ευρώπη και με τους ίδιους όρους και εκτός από την προστασία εντομένων και τα ηθικοπλαστικής φύσεως θέματα, αυτό που παίζει ρόλο κυρίως είναι η ασφάλεια. Κοιτάξτε, αυτά τα αεροσκάφη ε, όταν χρησιμοποιούνται βεβαίω και είναι ακριβά και για να κατασκευαστούν και για να τα αγοράσει κανείς. Και όταν κανείς ε, παίζει με αυτά, προφανώς δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ασφάλεια, δεν θέλει να επενδύσει σε αυτά. Όμω, Όμως ξέρετε και αυτά τα αεροσκάφη του μοντελισμού παρεμποδίζουν την ε, πολιτική αεροπορία, το πτυτικό έργο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν κάποιες εγγυήσεις, κάποιες ρυθμίσεις. Εντάξει, ό,τι θέλει να πετάει, να πετάει στον αέρα ε, και βέβαια και όλα τα άλλα υπτάμενα που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει, τα μπαλόνια και όλα τα διάφορα τα αερόστατα, αλλά εκείνο που παίζει ρόλο είναι να υπάρχει ένα αυστηρό σύστημα όπου θα μπορεί κανείς να διασφαλίσει συχνότητες για να μην προκύπτουν συγκρούσεις. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα, γιατί ξέρετε αυτό δεν αφορά μόνο τα μη παντρωμένα σκάφη, αφορά και τα μικρά αεροσκάφη. Επαναλαμβάνω την αρχή μου. Ό,τι μπορεί να πετάξει, να πετάει στον εναέριο χώρο, αλλά να μην υπάρχει ο κίνδυνος συντριβής, να αλληλοαναγνωρίζονται. Και αυτό αφορά και τα μικρά, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που και αυτά μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά. Η Γενική Διεύθυνση MOVE έχει τώρα το λόγο και ίσως μπορείτε και εσείς αν θέλετε να μιλήσετε για το πακέτο της αεροπλοίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Τζάκη και ευχαριστώ και όλους όσους πήραν το λόγο. Να πούμε και εμείς ορισμένα πράγματα πριν από δύο μήνες συζητήσαμε για πρώτη φορά την έκθεση αυτή και σημειώνω με χαρά ότι ήσασταν πάρα πολύ δραστήριοι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών σας. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες προκαταρτικές παρατηρήσεις πριν σχολιάσω τις συγκεκριμένες τροπολογίες. Νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση επίγοντος. Ε, η βιομηχανία και τα κράτη-μέλη ζητούν ε, κοινού κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εκτιμά την πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής σας, την πολύ καλή συνεργασία των σκιωδών εισηγητών και των διαφόρων πολιτικών ομάδων για να υπάρξει μια κοινή θέση πιο σημαντικές τροπολογίες τώρα. Το geofencing και η ανίσχυση των ε, drones ε, που είναι μέτρα ασφαλείας θα βελτιώσουν όχι μόνο την ασφάλεια αλλά θα βοηθήσουν ε, την αστυνομία και τις, τις αρχές προστασίας δεδομένων να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Είναι σημαντικό να υπάρχει κοινό πλαίσιο για όλα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ανεξαρτήτως της χρήσης τους. Γι' αυτό ε, η ε, τροπολογία 74 που είναι, αφορά την άρση του ορίου των 150 κιλών είναι πάρα πολύ ε, σημαντική. Μία πολύ ευρύτερη προσέγγιση η οποία θα είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Είναι επίσης πολύ σημαντική, γι' αυτό ο Τζάρους, οι κανονιστικές αρχές των μη επανδρομένων συστημάτων είναι πολύ σημαντικός φορέα. Είναι σημαντικό να συμμετέχει η ΕΑΖΑ ε, ώστε οι διεθνείς διατάξεις να είναι δεσμευτικοί κανόνες ε, με ε, τον κατάλληλο τρόπο. Συμβαστικές τροπολογίες 5 με 6 βρίσκουν πολύ καλή ισορροπία μεταξύ των διαδικασιών ΕΑΖΑ και Τζάρους και τονίζουν τη συμπληρωματικότητα. Τρίτον, τα, τα drones μπορούν να προβούν σε πολλές επιχειρήσεις μακριάς, μακράς εμβέλειας που δεν ε, μπορούσε να γίνει με, τις, ε, με, με άλλα μέσα στην πολιτική αεροπορία και υπάρχουν χαμηλού κινδύνου επιχειρήσεις ε, με, μέχρι επιχειρήσεις που έχουν την ίδια σημασία με επανδρομένα αεροσκάφη. Συμφωνούμε λοιπόν με ε, την αλλαγή που προτείνει η ε, τροπολογία 7. Δεν έχει σημασία κατά πόσο μιλάμε για εμπορική, επαγγελματική ή ε, χρήση για λόγους αναψυχής των συγκεκριμένων αεροσκαφών. Πρέπει οι κανόνες να, να παρέχουν ένα πλαίσιο προστασίας για τους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που τίθενται. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες ε, συγκεκριμένοι κανόνες όπως η ανείχνευση των drones ή το G-fencing ε, ελπίζουμε και συμφωνούμε με τέτοιου είδους μέτρα, όπως αυτά που προτείνονται στη συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 8. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκτιμά όλος ιδιαίτερο στην έκθεση ε, αυτή, η ΕΑΖΑ κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών δρομολόγησε για τα μικρότερα drones μία διαβούλευση και οι υπηρεσίες μου δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά για το είδος των drones που θα συμμετέχει σε αυτό το πακέτο, κάτι το οποίο θα εγκριθεί πριν από το τέλος του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό απαντά και στην ερώτηση που, έχουν, που έχετε θέσει πολύ εξημών, δηλαδή τι πρόκειται να κάνει η συγκεκριμένη επιτροπή. Θέλουμε να βελτιώσουμε την πιστοποίηση, αλλά πρέπει να δούμε και άλλους τομείς και όπως είπα και προηγουμένως δεν έχουμε χρόνο, επομένως οι προτάσεις πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι το τέλος του έτους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα η κυρία Τζάκι Φώστερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλια όχι μόνο από τους κοιόδης εισηγητές αλλά και από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλια της. Μόνο μερικά σημεία θα ήθελα να ε, θέσω. Είναι κατανοητό ότι μπορεί να υπάρχει ανησυχία. Ε, η κυρία Αγνωτό ε, ανέφερε και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε, πολύ βασικό όταν μίλησε για την έμφαση στις εθνικές αρχές που ασχολούνται με το θέμα αυτό, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είπε και άλλοι συνάδελφοι, είναι πολύ ευρύτερο από το εθνικό γιατί χρησιμοποιούμε τον αέριο χώρο και βεβαίως θέλουμε οι εθνικές κυβερνήσεις, αναμένουμε να έχουν κανόνες ε, ε, Κυριαρχία όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά πρόκειται για ένα διεθνές παγκόσμιο εγχείρημα, ε, το οποίο ε, ελπίζω να το κατανοείτε και να σας ησυχάζει. Κάτι το οποίο είπατε Ευρω... Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των επενδύσεων. Εμεί δεν ζητήσαμε ποσό, εμείς είπαμε, έχουμε τον ορίζοντα 2020, έχουμε το ΣΕΖΑΡ, γιατί πρόκειται για έναν τομέα εξελισσόμενο, αναπτυσσόμενο, Είχατε πει 30 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο το οποίο θα ε, παρασχεθεί για επενδύσεις. Ε, πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτο. Σας ευχαριστούμε πολύ παρά το γεγονός ότι δεν ξέρω από πού ακριβώς προέρχεται αυτό το ποσό. Δύο ακόμη ε, σχόλια. Υπάρχει ακριβώς ιδιαίτερη έμφαση στη διάκριση μεταξύ επαγγελματικής χρήσης και χρήσης για λόγους αναψυχή. Εμείς δεν θέλουμε να δέσουμε χειροπόδαρα έναν άνθρωπο ο οποίος για λόγους αναψυχή θέλει να χρησιμοποιήσει ένα ντρόουν. Όμως εφόσον χρησιμοποιεί ένα αέριο χώρο αυτό πρέπει να το παντρέψουμε κάπως με ευρύτερες χρήσεις και ευρύτερα ε, αεροσκάφη. Γι' αυτό ακριβώς έπρεπε να το γράψουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Το geofencing ε, και το ε, βλέπε και απόφευγε, detect and avoid. σε 36.000 πόδια ύψος ε, ο, το τελευταίο που θέλουμε είναι να υπάρχουν διάφορα μικρά αεροσκάφη τα οποία θα μπαίνουν ε, ε, στην ε, διαδρομή μας και θα την παρεμποδίζουν. Είναι φυσικό, έχουμε την τεχνολογία να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Όλα αυτά τα μέτρα, τα τεχνολογικά που μπορούν να ληφθούν, πρέπει να ληφθούν ώστε να μπορέσουμε να προστατευτούμε και εν πτήση αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είπατε. Ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αν θέλετε το απόγευμα να, το δούμε μαζί και να δούμε πώς, μπορούμε να, ε, ε, πώς μπορεί να συμπεριληφθεί στις συζητήσει μας ε, αύριο το πρωί, ίσως όταν θα γίνει ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους. Νομίζω ότι ήταν ε, μια εξαιρετική δουλειά. Ε, στην οποία συμμετείχαμε όλοι και ελπίζω ότι θα πάει εξίσου καλά και αύριο ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αύριο ψηφίζουμε και πάλι για την έκθεση αυτή στις 9 η ώρα ακριβώς. Έτσι. Ωραία. Επόμενο θέμα τώρα στην ημερήσια διάταξη. Νέε προκλήσει και έννοιε για την πρόοδο του τουρισμού στην Ευρώπη. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ιζαμπέλα Ντεμόντε και βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που στέκονται όρθιοι Καθίστε εκεί που είναι ε, οι πράσινες ε, ταμπελίτσες των αναπληρωτών για να μπορείτε να ακούτε και τη διερμηνία, αν επιθυμείτε. Εκτός αν έρθουν οι βουλευτές οι οποίοι φυσικά προηγούνται. Αλλά για να μην έχουμε κενά να δεν υπάρχει λόγος να στέκεστε όρθιοι και να μην ακούτε και τη διερμηνία.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 Σα eh, eh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα λοιπόν έχουμε να εξετάσουμε τις ε, τροπολογίες ε, περίπου 150. Μιλάμε για πολύ μεγάλη συνεισφορά εκ μέρους των ε, συναντέλφων. Και θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους ε, που με βοήθησαν, επίσης όλους τους συναδέλφους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν και αυτοί. Ε, επίσης, ε, θέλω να πω το εξής, όλες αυτές οι τροπολογίες επέτρεψαν στο να καταλήξουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις Επιτροπές της Εσωτερικής Αγοράς, του Πολιτισμού και της Παιδείας, γιατί με τη δική τους την άποψη συνέβαλαν βοήθησαν στη σύνταξη των συμβασικών προτάσεων όπου ελήφθησαν υπόψη οι δικές τους οι απόψεις. Νομίζω ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι καταλήξαμε σε συμβιβασμούς ε, γιατί είμαι πεπισμένη ότι οι δραστηριότητες μας στον τομέα του τουρισμού δεν πρέπει να έχουν πολιτικά σύνορα. Ε, θα πρέπει να φορούν όλες τις ομάδες. Επίσης θεωρώ ότι αυτή η πρόταση πρωτοβουλίας θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική αν τελικά κατορτώσουμε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Όλες λοιπόν αυτές οι συμβαστικές προτάσεις έδωσαν μια όθηση σε τρεις τομείς που είναι ο πολιτισμός, εκεί γίνεται λόγος ε, για τη διατήρηση της πολιτικής κληρονομιάς, ε, της προστασίας της UNESCO. Αυτό που επίσης ε, προβάλλεται ιδιαίτερα είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πέρα από, την, ε, από όλα αυτά υπάρχει και η χρήση της ε, πύλης Visit Europe Έχουμε και την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αυτό κυρίως για να προωθείται η απασχόληση στους ε, νέους ε, Ευρωπαίους και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου, κυρίως ε, κάτω από το πρίσμα της ανεργίας, διότι η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους. Κατόπιν υπάρχει το θέμα του προϋπολογισμού. Εκεί πάρα πολλοί συνάδελφοι επισήμαναν ο τουρισμός να έχει την δική του την γραμμή στον προϋπολογισμό αντί να είναι διάσπαρτος σε πολλά άλλα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται ε, και μέσω αυτών χρηματοδοτείται και ο τουρισμός να υπάρχει επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια, να μεταφράζονται τα κείμενα σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Αυτό είναι κάτι που έρχεται και επανέρχεται, δηλαδή ότι η μετάφραση είναι πολύ σημαντική και είναι σημαντικό να υπάρχει μετάφραση σε περισσότερες γλώσσες. Οι συμβαστικές προτάσεις αφορούν και στην αναγκαιότητα να υπάρχουν ειδικά προϊόντα για να αυξάνονται οι τουριστικές ροές. Δηλαδή να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο είδος του τουρισμού που θέλουμε να ενισχύσουμε. Και πρέπει και πάλι να ενισχυθούν οι απομακρυσμένες ε, περιοχές, ε, οι ε, ορεινές, οι περιφερειοποιημένες και όλα αυτά γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν προαχθούν αυτές οι περιοχές αυτό δεν ευνοεί την οικονομία ούτε τη σταθερότητα να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους πιο ηλικιωμένους, ε, σε άτομα με αναπηρία και να ενδιαφερόμαστε για έναν τουρισμό για όλους. Αυτή εξάλλου είναι και η άποψη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Όσον αφορά τώρα το Brand Europe, αυτή την ε, ε, εμπορική ονομασία, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη συνεργασία ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως στην πρόσβαση των κονδυλίων. Ε, Αϊφόρος και βιώσιμος ε, τουρισμός. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε κάποια ιδιαίτερα, ιδιαίτερους κύκλους ε, μαθημάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανακύκλωση, για τη θρησκεία, για οτιδήποτε. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο. Θα πρέπει κανείς να γνωρίζει τις διάφορες προσεγγίσεις, αλλά και εδώ καταλήξαμε σε μία συμφωνία και υπογραμμίζουμε κυρίως το πόσο σημαντικό είναι να πριν προκύψει κάποιος κανισμός, γιατί αυτή τη στιγμή διάφορα κράτη-μέλη λειτουργούν αυτόνομα, αυτό που έχει σημασία είναι να λαμβάνεται υπόψη η προστασία των καταναλωτών ε, και η ψηφιοποίηση κυρίως ε, για την διάδοση των, ε, της ευρυζωνικότητας στις πιο απομακρυσμένες ε, περιοχές. Δεν κατέστη βέβαια δυνατό να συμπεριλάβω όλους, όλες τις τροπολογίες του συμβασμού Υπάρχουν όμως πολύ σημαντικές προτάσεις που κατατέθηκαν. Εμένα με ενδιέφερε να διατηρήσω μια γραμμή και Νομίζω ότι πάνω σε αυτό μπορούμε αν θέλετε να συζητήσουμε και αύριο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα δούμε τι θα παραμείνει και τι όχι. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι σε τελική ανάλυση πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εμπειρία. Ε, οι συνάδελφοι με βοήθησαν πάρα πολύ και ελπίζω αύριο ε, και με τις ερωταπαντήσεις θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Κλάουδια Μοντέρο Νταγκογιά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για ε, όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει για το συγκεκριμένο έγγραφο. Θα ήθελα επίσης να την ευχαριστήσω και για τις εξηγήσει που μόλις μας έδωσε προφορικά. Ήταν ε, συνενετική ε, η συνεργασία μας. Ήταν πάνω από 350 οι τροπολογίες που κατέληξαν σε 21 συμβαστικές. Και τελικά το κείμενο φέρει τη σφραγίδα όλων μας. Έχουμε καλύψει πολλά σημεία και πολλές πτυχές, τα είπε και η συγκήτρια. Η συμμετοχική οικονομία, η ψηφιοποίηση, ε, καλύπτονται το θέμα του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος της μάρκας Ευρώπη ε, και ε, της προώθησης. Αυτό το τελευταίο θέλω να το τονίσω γιατί όταν μιλούμε για τον τουρισμό το 90% των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις ή ε, μεσές και χρειάζεται να βελτιώνεται η χρηματοδότησή τους. Θα ήθελα να εμφερθώ και σε άλλα σημεία που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Η γαλάζια οικονομία, ο τουρισμός σε παραθαλάσσιες περιοχές χρειάζεται ένα πρόγραμμα δράσης. Πέρα από τις 14 δράσεις που ήδη έχουν ε, προβλεφθεί για την προστασία του παραθαλάσσιου τουρισμού, όπου εργάζονται πάνω από 3 εκατομμύρια ε, πολίτες και είναι από τις σημαντικότερες ε, δραστηριότητες στην Ευρώπη. Ένα μεγάλο τμήμα των επιχειρήσεων πάνω στην Ευρώπη ε, αποσκοπεί εκεί. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα στη θάλασσα δεν είναι μόνο η παραλία και ο ήλιος, ε, αλλά και διαφοροποιημένα προϊόντα, αφήση, γαστρονομία, αθλητισμός, κρουαζιέρες, ε, θαλάσσια αθλήματα και τα λοιπά. Θα πρέπει να έχουμε μια ε, διακρατική συνεργασία, ε, βέβαια και σε τοπικό επίπεδο μεταξύ διαφορών ε, κρατών. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι παντού η ίδια η διάρκεια της σεζόν στις παραθαλάσσιες περιοχές. Επίσης, κάτι άλλο που λέει η έκθεση είναι η προσβασιμότητα. Η προσβασιμότητα των χερσαίων και των ισιωτικών περιοχών. Αυτό έχει να κάνει ε, με τις συγκοινωνίες και τις συνδέσεις. Ε, έχουμε τις ακτοπλοϊκές, τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Ε, αυτά τα παραθαλάσσια μέρη και τα νησιά είναι κυρίως τουριστικά. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρχει καλή πρόσβαση. Ε, διαφοροποιημένα όμως δεν μπορούμε να έχουμε νέους κανόνες οτιδήποτε ισχύει ε, παντού να ισχύει και για τις απομακρυσμένες περιφέρειες και για τα νησιά μας. Χρειάζεται μια σαφής στρατηγική με καλή προετοιμασία και μεθοδική και ε, για την ανάπτυξη προϊόντων και διακρατικών υπηρεσιών που παρέχονται. Και αυτή η στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει όλο τον τομέα και το δημόσιο και τον ιδιωτικό. Να αναπτυχθεί αυτή η μάρκα Ευρώπη, αλλά με ιδιωτικές επενδύσεις. Γιατί δεν μπορούμε να τα ζητάμε όλα από το κράτος ή να εξαρτώμαστε πάντα από κρατικές επενδύσεις. Κοιτάξτε μερικά παραδείγματα. Και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένε Πολιτείες και στον Καναδά, ε, έχουν ένα brand name και για τον τουρισμό. Και εμεί θα πρέπει να έχουμε αυτή τη στρατηγική για να προσελκύσουμε και καινούριου τουρίστε σε άλλε περιφέρειε, πέρα από τι κλασικέ γνωστέ ε, ε, τουριστικέ περιοχέ. Και τέλο, χρειάζονται υποστήριξη και οι νέοι. 45% των εργαζομένων στον τουρισμό είναι νέοι. Η συγγήτρια Ισαμπέλα το είπε προηγουμένως. Περί δηλαδή, αυτού πρόκειται. Θέσεις εργασίας για νέους ιδιαίτερα και γι' αυτό θα πρέπει επιγόντως να ασχοληθούμε με το θέμα. Αυτά. Και γι' αυτό χρειάζεται πάντα ειδική χρηματοδότηση και ειδική γραμμή στον προπολογισμό για τον τουρισμό. Γιατί ο τομέας αυτός δεν θα πρέπει να είναι στο περιθώριο το αποπέδι είναι τεράστιο, το δυναμικό μπορεί να δημιουργήσει πλούτο σε διάφορα κράτη-μέλη και υπάρχει και τεράστια δυνατότητα για νέες θέσεις εργασίας. Το κείμενο που θα ψηφίσουμε αύριο νομίζω είναι μια εξαιρετική αφετηρία που μπορεί να μετεξελιχθεί και να βελτιωθεί για να εφαρμόσουμε τις απαραίτητες εκείνες δράσεις ε, που χρειαζόμαστε για τον τουρισμό και θα βελτιώσει την κατάσταση στην Ευρώπη γενικά. Ευχαριστώ. Ο Γιώργος Ράντους. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο λέγοντας ότι η κυρία Ντεμόντε είχε, ε, έκανε εξαιρετική δουλειά. Ε, να τη συγχαρώ λοιπόν για την έκθεσή σας και κατά την προετοιμασία ήταν ε, πάρα πολύ καλή δουλειά. Ένα θέμα μόνο θα ήθελα να θέσω που είναι το θέμα του συντονισμού. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, έχετε, δεν έχει νομοθετικές εξουσίες ε, για τον τουρισμό και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές μιλάμε ε, σε αυτή την έκθεση για το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων παικτών ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το βασικό φορέα. Αν αυτά τα μοντέλα συντονισμού ε, είναι καλά. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και γι' αυτό ακριβώς εκ μέρους ε, της ομάδας των φιλελευθέρων εγώ θα ήθελα να προτείνω μια τροπολογία ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεύρει τρόπους αποτελεσματικού συντονισμού και συνεργασίας ε, στον τομέα του τουρισμού. Και σας καλώ εσάς αγαπητοί συνάδελφοι να υποστηρίξετε την πρόταση αυτή της ομάδας μου. Ευχαριστώ η Μαρία Κίλωνεν. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτά που ήδη έχουν υποθεί. Ήταν πολύ καλά τα σχόλια και δεν χρειάζεται να προσθέσω πολλά. Το μόνο που έχω να πω είναι θέλω να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια και τους εισηγητές για την εξαιρετική τους ε, δουλειά εδώ, αλλά θα ήθελα να τονίσω και κάτι ακόμα, μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στον τουρισμό και μάλιστα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Θεώρηση, θεώρηση και ξανά θεώρηση, διαβατηρίων εννοώ. Η πολιτική μας για τις θεωρήσεις είναι ένα τεράστιο εμπόδιο και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι κάνουν η Αυστραλία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλοι ε, εταίροι μας ε, στις θεωρήσεις διαβατηρίων για να ε, προσελκύουν ας πούμε τουρίστες από την Ασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το είχαμε πει και εδώ στην Επιτροπή μας το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα, όντως έχει μεγάλη σημασία. Το λόγο τώρα έχει η Καριμά Ντελή. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος ε, ε, Jill Evans ε, δεν είναι εδώ και μου ζήτησε εκ μέρους της να σας συγχαρώ για την δουλειά σας. Πάρα πολύ καλή συνεργασία που μας επέτρεψε να έχουμε τροπολογίες που σε μεγάλο βαθμό είναι αρκετά θετικές για την οικολογία. Ναι, ε, ναι στον τουρισμό, δεν τον μεταχειριζόμαστε σήμερα όπως το κάναμε ε, πριν από κάποια χρόνια. Μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό τώρα, ζητάμε περισσότερη κινητικότητα, ε, προστασία της κληρονομιάς και να υπάρξει βέβαια ευαισθησία από τον τουρισμό αυτό προς τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή με αναπηρία τονίσατε, το είπατε κιόλας, ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία ειδικότερα στις ε, ορεινές ή παράκτιες περιοχές. Είναι αλήθεια όμως ότι η έννοια της κλιματικής αλλαγής πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση γιατί η κλιματική αλλαγή σε σχέση με τις περιοχές αυτές είναι κάτι το πολύ σημαντικό Πρέπει λοιπόν να, γίνει, να υπάρξει ε, σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά αυτή η έκθεση ένα πολύ καλό παράδειγμα ε, του, δε έπρεπε, του τι δεν θα έπρεπε να ε, κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι εθνική αρμοδιότητα ο τουρισμός ε, γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά. Ε, για παράδειγμα στη Σουηδία υπάρχει το θέμα της πολύ όμορφης φύσης. Στην Ισπανία πάει κανείς για τον ήλιο και τις παραλίες. Είναι λοιπόν διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του τουρισμού ανάλογα με τη χώρα. Ε, ο, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πολίτες κάνουν την εμπιστοσύνη τους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο και ίσως θα έπρεπε πριν αρχίσουμε να πλησιάζουμε τέτοιου είδους τομείς να το σκεφτόμαστε και αυτό. Η κυρία Μαρή Κριστίνα Αρνουτού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία εισηγήτρια Ντεμόντε για την εργασία της αυτή. Βεβαίως, ο τουρισμός είναι μείζον κλάδος της οικονομίας των ευρωπαϊκών κρατών και βεβαίως και στο μέλλον ο αριθμός των τουριστών θα αυξηθεί. Αλλά για να ανταποκριθούμε σε αυτή την αύξηση θεωρείται κυρία η ότι η ψηφιοποίηση και ε, η ε, οικονομία η συμμετοχική είναι βασικές λύσεις. Ε, δεν λαμβάνεται υπόψη. Εντάξει, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, αλλά δεν είναι προτεραιότητα. Η βασική όμως πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τουρισμός και θα αντιμετωπίσει σίγουρα και τα επόμενα χρόνια είναι τελείως διαφορετική. Πρόκειται για την αύξηση της ανασφάλειας. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό αυτό το πρόβλημα που αφορά άμεσα και πλήττει την τουριστική βιομηχανία. Και αν δεν το λύσουμε γρήγορα φοβούμε ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Οι τουρίστε πηγαίνουν σε χώρε που αισθάνονται ασφαλείς και εξασφαλίζεται και η σωματική του ακαιρεότητα και η ηλική του. Στην ασφάλεια όμω, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι όλο και περισσότερο ε, μειώνεται η ασφάλεια στην Ευρώπη και πρέπει να τον αναγνωρίσετε. Και ε, με αυτά τα κύματα μεταναστών που έχουμε δεν βελτιώνεται. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Πριν από δύο χρόνια η ασφάλεια στο Παρίσι, ήταν, η ανασφάλεια μάλλον, ε, ήταν ε, μια τέτοια μάστιγα που έκανε διάβημα η Κινέζικη Πρεσβεία. Τον Απρίλιο του 2013 έκαναν απεργία οι φύλακες ε, στο Λούβρο γιατί αυξήθηκαν πάρα πολύ οι πορτοφολάκιδες. Επίσης τα πολυτελή καταστήματα διαμαρτύρονται. Ε, την περασμένη εβδομάδα ε, κοντά στην, ε, στο καθεδρικό Νότρο Ντάμ μια γυναίκα έβγαζε χρήματα και της επιτέθηκαν η Ρομ και το έγραψε και Daily Mail αυτό. Στην Νίκη από όπου κατάγομαι είναι πάρα πολλοί τουρίστες και πάρα πολύ συχνά ο τύπος της περιοχής εκεί αναφέρει επεισόδια μια Ιρλανδή που την έδιραν και την έκαψαν, και από άλλα, από τη Σουηδία ας πούμε, μια ε, τουρίστρια η οποία ξυλοκοπήθηκε και ε, στη συνέχεια ε, Υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και ο δράστης 24 χρονών Ρουμάνος άστεγος είχε επιτεθεί σε ένα πάρκο και είχε βιάσει μία Ελβετίδα τουρίστρια. Όλα αυτά λοιπόν ε, ε, και βλέπουμε να δηλώνουν τουρίστες ότι δεν θα ξαναπατήσουν το πόδι τους στην Νίκαια. Ε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ε, φυσικό να συμβαίνουν και ε, η ανασφάλεια επίσης στα λεωφορεία και τα τουριστικά λεωφορεία τους κατακλέβουν στο μετρό, στον προαστιακό, τους κλέβουν τα πράγματα, τα πορτοφόλια, ε, τους χτυπάνε και ακριβώς οι τουρίστες είναι ένας στόχος για να μην γίνει λόγος και για ε, τις τρομοκρατικές επιθέσεις στα τρένα. Με τέτοια κακή διαφήμιση δεν είναι απορίας άξιο να πέφτει το Παρίσι στις διεθνείς καταστάσεις ως προορισμός. Όλα αυτά κινδυνεύουν να ε, φέρουν σε μόνιμη αναταραχή την κατάσταση και στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα λοιπόν, η έλλειψη ασφάλειας και φοβούμε ότι τα επόμενα έτη θα επιδεινωθεί. Άρα αυτό το σημαντικό και σοβαρό θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί και είναι μια νέα πρόκληση. Αυτή είναι νέα πρόκληση και ιδιαίτερα κεφαλαιόδου σημασία θα πρέπει δεν να αναγράφεται στην πρόταση αυτή ψηφίσματος. Μπορεί να μην ε, σας ενδιαφέρει όλους τους παρόντες εδώ, αλλά πιστέψτε με ανησυχεί πάρα πολύ. Έχει θορυβήσει τους Γάλλους ε, πολίτες που εδώ εκπροσωπώ. Θέλω λοιπόν, είναι σημαντικό να εγγραφεί ε, αυτό το θέμα ως σημαντική πρόκληση για το τουριστικό τομέα σήμερα και έκανα και μια τροπολογία σχετικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Κιστίνε Μάισνα. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ σύντομα για να απαντήσω σε συνάδελφο Λουντ Γκριν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό. Βεβαίω και ο τουρισμό γενικά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Μόνο που αν θέλουμε να προβάλλουμε την Ευρώπη ω υπαριθμόν ένα τουριστικό στόχο στον κόσμο, ε, πρέπει να το προσπαθήσουμε και Ξέρετε, αυτό δεν είναι ακόμα νόμος, μια έκθεση είναι. Βεβαίως και αν υπάρξει νόμος από την Κομισιόν για τον τουρισμό, τότε θα το λάβει αυτό υπόψη του το Κοινοβούλιο και δεν πρέπει και να υπερβάλλουμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ το να ζητήσουμε τώρα ε, έναν τουριστικό φορέα. Ε, καλύτερα να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε μια πλατφόρμα. Ε, και κάτι άλλο θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές ε, στον ε, τουρισμό ε, υπάρχουν πολλές οικονομικές δυνάμεις. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε όλα αυτά να τα προάγουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μία τελευταία παρατήρηση. Υπάρχει μία τροπολογία του, τον Άλντε για το ticketing και από ό,τι άκουσα αυτό δεν το εγκρίνουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Εγώ δεν λέω στις πολιτικές ομάδες τι να ψηφίσουν, αλλά πιστεύω ότι το integrated ticketing αυτό έχει σχέση με τον τουρισμό. Ε, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το ολοκληρωμένο εισιτήριο, να μπορώ να βάλω στο ίντερνετ που θέλω να πάω, από πού φεύγω και να έχω έτσι ένα πλήρες εισιτήριο με όλα τα μέσα μεταφορών. Η Λούσι Άντερσον έχει το λόγο. Συγχαίρω την εισηγήτρια και τους σκιώτης για την έκθεσή τους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανασφάλειες στην Ευρώπη, να προβάλλουμε τη σημασία της Ευρώπης ως ε, βασικό ε, τουριστικό προορισμό τη σημασία του τουρισμού για την οικονομία. Νομίζω ότι όλε αυτέ οι τροπολογίε είναι ιδιαίτερα θετικέ. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά που ελέγχθησαν για την κρίση σχετικά με την ασφάλεια των μεταφορών. Εντάξει, υπάρχουν θέματα που εξετάζονται, εκεί έχετε δίκιο. Νομίζω όμω ότι όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε μέσα σε μία προοπτική. Και υπάρχει ένα τομέα που είναι σημαντικό ε, για την ασφάλεια του τουρισμού. Αυτός έχει σχέση με τα καταλήμματα ε, κυρίως ε, αν θέλετε και με την ασφάλεια από πυρκαγιές, ε, τη μη έκκληση μονοξιδίου του άνθρακα. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Έχει φτάσει λοιπόν η χρονική στιγμή να ληφθούν μέτρα. Οι συνάδελφοί μου από την αντιπροσωπεία των εργατικών και του Ρωμένου Βασιλείου ανησυχούν πάρα πολύ ε, σχετικά με όλα αυτά που σας είπα γιατί υπάρχει και μια σχετική περίπτωση ενός Βρετανού πολίτη και πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ε, επίσης, όσον αφορά την ε, πρόσβαση και την προσπελασιμότητα για άτομα με ειδικέ ανάγκες. Ε, αυτό επίσης είναι ένα θέμα που κατά την άποψή μου πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η κυρία Σαγιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ και την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για την έκθεση αυτή. Είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη για ένα από τους κλάδους της οικονομίας που είναι πολλά υποσχόμενη και που ε, υπόσχεται και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Αυτό που θέλω να πω μόνο είναι να αναφερθώ σε κάποιες από τις προκλήσεις που έχουμε. Και αυτές έχουν να ε, κάνουν με τις νέες τεχνολογίες, τις, τις πολύ τελευταίες ε, και ένα τομέα όπως είναι ο τουρισμός όπου υπήρξε ρύθμιση για όλους τους συμμετέχοντες, υγιεινή, ασφάλεια, δικαιώματα εργαζομένων κτλ. Ε, έχει εποχιακό χαρακτήρα αυτός ο κλάδος και έχουν και κάποια συγγραφή υποχρεώσεων. Και απ' την άλλη βλέπουμε διάφορες πλατφόρμες, μοντέρνες, ε, για τους νέους, ελκυστικές, όπου ε, κάποιος παρέχει μια υπηρεσία, ένας ιδιώτης και όλος ο χρήστης θεωρεί ότι θα κάνει οικονομία ε, και δεν θα έχει διάφορες υποχρεώσεις και βλέπουμε στη Βαρκελόνη τι γίνεται ας πούμε αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου ένας κλάδος ο οποίος στην Ευρώπη έχει παράδοση, ιστορία ε, ρύθμιση, πλαίσιο και λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και με ένα κύρος και μία έγλη, ε, όλα αυτά ε, ανατρέπονται στο βωμό της μοντέρνας προσέγγισης και θέλουν να παρακάψουν όλες αυτές τις ιστορικές δεσμεύσεις και ρυθμίσεις μετά από όλα αυτά τα χρόνια στο βωμό του σύγχρονου και του μοντέρνου. Μα υπάρχουν θέματα ασφάλειας, ε, απάτης, να μην κλέβεις τον άλλον όταν έρχεται και ε, επισκέπτεται τον τόπο σου. Ε, είναι ζητήματα συγκεκριμένα αυτά. Καλή είναι η μοντέρνα εποχή, αλλά να μην καταστρέψουμε ολόκληρους κλάδους της οικονομίας, έτσι δεν είναι. Σας είπα, έχει κάνει τεράστια προσπάθεια ο κλάδος για να ψηφιοποιηθεί, να προσθέσει ε, πιο κοντινές στο χρήστη φόρμουλες, πλατφόρμες, ηλεκτρονικά. Αλλά αυτό είναι ένα. Μέχρι να τα καταργήσουμε όλα και να τα ισοπεδώσουμε όλα, τα κοινωνικά, τα δικαιώματα, τα πλαίσια κτλ. Κάπου χρειάζεται να τραβήξει μια κόκκινη γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ είχα βάλει το όνομά μου και θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος Λούντκριν. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ο τουρισμός δεν είναι εθνική υπόθεση. Ακούω, ας πούμε, στη Φινλανδία, οι δυτικοί Φινλανδοί δεν καταλαβαίνουν ε, κατά πόσο υπάρχουν τρελοί Ευρωπαίοι που πάνε στην Ανατολική Φινλανδία και κάνουν διακοπές. Και οι νότιοι Σουηδοί δεν μπορούν καν να φανταστούν ότι η Βόρεια Σουηδία είναι περιοχή τουρισμού. Γι' αυτό, να, ξέρετε, οι περιφέρειες πρέπει να συνεργαστούν και μερικές φορές είναι σωστό να συνεργάζονται διασυνοριακά στην ε, Ευρώπη. Το κάναμε αυτό, την στρατηγική της ε, Βαλτικής θάλασσας και αυτοί εκμεταλλεύονται τη Βαλτική θάλασσα όλοι από μαζί, όχι ο ένας ενάντια στον άλλο. Αυτό είναι πολύ επιτυχημένο. Και στο Δούναβι και εκεί συμμετέχουν όχι μόνο οι παράκτης χώρες, αλλά και αυτές που είναι στα υπηρετικά, ε, γιατί μπορούν να προβάλλουν το Δούναβι και να τον εκμεταλλευτούν και σε επίπεδο μουσικής, όλα αυτά να τα προβάλλουν σε τουριστικό επίπεδο και αυτό είναι ευρωπαϊκό καθήκον. Βεβαίως ο τουρισμός είναι κάτι περιφερειακό, κάτι εθνικό αλλά και κάτι ευρωπαϊκό και νομίζω αυτό πρέπει να το τηρήσουμε. Αυτό ήθελα να πω και δίνω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ πλήρης έκθεση της κυρίας Δεμόντε. Νομίζω ότι ε, πραγματεύεται τις βασικές προκλήσεις του τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ε, τις ε, συστάσεις. Θα ήθελα επίση να σας ενημερώσω ότι θα υπάρξει ένα φόρουμ αυτή την εβδομάδα στο Λουξεμβούργο υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για σημαντικά θέματα όπω ε, η προώθηση του τουρισμού, ε, η πρόκληση του, της, ε, της χρήσης των ψηφιακών πλατφορμών. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομο ήταν. Πραγματικά εκπλαγήκαμε όλοι και τώρα έχει η συγγήτρια το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις ε, παρεμβάσεις. Ευχαριστώ τους και ηγητέ, του συναδέλφους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, νομίζω ότι ε, συμμερίζονται όλοι και συμφωνούν με τους συμβασμούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους κυρίως διότι ανέφεραν το θέμα της νεανικής ανεργίας, το πόσο ε, σημαντικό είναι όλοι οι τομείς του τουρισμού να προσφέρουν απασχόληση. Τώρα, είναι απαραίτητο πράγματι να υπάρχει συντονισμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται και σε μία τροπολογία και είναι αλήθεια ότι ο τουρισμός είναι εθνική αρμοδιότητα, από την άλλη όμως θα πρέπει να προβάλλουμε ένα εμπορικό σήμα, ένα μπραντ που να είναι υπερεθνικό κατόπιν τούτου θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μία οργάνωση που να είναι συνεπής με όλα αυτά που αναφέραμε. Τώρα για τις θεωρήσεις. Είχαμε τοποθετηθεί και είναι απολύτως απαραίτητο να ακολουθήσουμε μία κατεύθυνση η οποία θα μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση και πέρα, και πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα τα θέματα τα κλιματικά ε, τα εξετάσαμε αυτά ε, στο πλαίσιο του Συμβασμού για την παράγραφο υπαριθμών 18 ε, και μάλιστα ασχοληθήκαμε και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι πιο απομακρυσμένες περιοχές είναι και οι πιο ευαίσθητες. Εξάλλου, αυτές είναι και πιο ευπαθείς και τροτές στις κλιματικές αλλαγές. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε και εκεί να παρέμβουμε, να παρέμβουμε λοιπόν στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί θεωρώ ότι εδώ μπορούν να υπάρξουν σημαντικές επενδύσεις. Όσον αφορά την ασφάλεια, ελέγχθησαν τα πιο σημαντικά θέματα. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που θέλω να πω είναι σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Αύριο θα ψηφίσουμε. Ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι απόλυτα ικανοποιητικό και έτσι λοιπόν ε, είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε να μιλάνε και άλλοι στην άλλη από αυτού του θέματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ψηφοφορία αύριο το πρωί ως και προχωράμε στην επόμενη έκθεση για τον τουρισμό επαναλαμβάνει ο πρόεδρος την ίδια έκθεση που μόλις τελειώσαμε. Λάθος. Βιώσιμη αστική κινητικότητα. Μα πώς είναι δυνατόν. Ναι, ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Ε, εντάξει. Ε, είπαμε, τελειώσαμε και αύριο είναι ψηφοφορία για να το εμπεδώσουμε. Ε, βιώσιμη αστική κινητικότητα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Καριμαντελή, στην οποία και δίνω αμέσω το λόγο μια στιγμή λίγο να αλλάξει η κατάσταση και να επανέλθει η προσοχή. glaube, jetzt παρακαλώ, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς, είναι σημαντικό, να ευχαριστήσω τους σκιώδης ηγητές για τη ε, δουλειά τους, οι οποίοι προσπαθούν ε, να καταλήξουμε σε τολμηρούς και ποιοτικού ε, συμβιβασμούς. 502 τροπολογίες, 50 τροπολογίες συμβιβαστικές που ακόμη τις συζητούμε αλλά νομίζω ότι με μεγάλα βήματα πλησιάζουμε ε, προς μία ε, στέρεη συμφωνία. Θα πρέπει η κινητικότητα να μην είναι αυτός σκοπός, αλλά να είναι ένας στόχος. 80% των πολιτών θα ζουν σε αστικά κέντρα ε, σύντομα. Πρέπει λοιπόν όλοι, ακόμη και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, να έχουν πρόσβαση στα πάντα, στο σχολείο, στη δουλειά, ε, στον πολιτισμό, στην αναψυχή, στην ε, υγεία. Παρ' όλα αυτά η αστική κινητικότητα είναι ένας περιορισμός ε, στην Ευρώπη. Η εξάρτηση από το αυτοκίνητο και από τα μποτιλιαρίσματα σημαίνουν ότι γίνονται όμοιροι μιας κακής κινητικότητας οι πολίτες. Μερικές φορές μάλιστα φτάνουμε σε εντελώς παράλογα πράγματα γιατί 50% των αστικών μεταφορών δεν υπερβαίνουν τα 5 χιλιόμετρα. Οπότε η φιλοδοξία της έκθεσής μου είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση του 21ου αιώνα. Μία ερώτηση ε, πώς μπορούμε να ε, βελτιώσουμε τη μετακίνησή μας. Υπάρχουν πάρα πολλά επίγοντα ζητήματα. Καταρχάς, το θέμα του κλίματος. Ε, η γεωργία και η βιομηχανία έχουν μειώσει ε, τις εκπομπές αερίων τους, αλλά οι μεταφορές από το 1990 έχουν αυξήσει κατά 30% τις εκπομπές τους είναι το 1 τέταρτο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου λόγω των οδικών μεταφορών κυρίω. Είναι σημαντικό να αντιστρέψουμε αυτή τη τάση αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιτύχει του στόχου που έχει ε, θέσει μέχρι το 2030 όσον αφορά τι εκπομπέ αερίων. Υπάρχει και μία, ένα, κάτι, κάτι, επίγον από απόψεως υγείας. Υπάρχουν εχμές ρήπανσης ε, που επηρεάζουν τους ε, πολίτες. Περίπου 4.000 θάνατοι κατέτος ε, οφείλονται στα ε, σωματίδια από τη ρήπανση που προκαλούν οι κινητήρες δίζελ σε μεγάλο βαθμό. Επομένως δεν πρέπει να, κολυσι, να κολυσιεργούμε. Ακόμα και ο ΙΕ το λέει από το 2050 η, η ρήπανση ατμοσφαιρική θα είναι ε, υπεύθυνη για το 1 πέμπτο των θανάτων, ε, ε, των θανάτων. Ε, πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να καταργήσουμε τους κινητήρες diesel. Εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να μου πούνε ότι δεν έκανα τίποτε και να με κατηγορήσουν στο μέλλον ότι δεν έκανα απολύτω τίποτε για να αντιστρέψω αυτή την κατάσταση. Κάτι άλλο είναι πολύ επίγον ε, η ζωή των ε, χρηστών του οδικού δικτύου. 38% των θανάτων ε, οφείλονται σε ε, οδικά ατυχήματα που συμβαίνουν στην πόλη, στα αστικά κέντρα. 25.845 νεκροί στα οδικά δίκτυα, περίπου 203.150 ε, το 2013 μόνο. Επομένως πρόκειται για μια κατάσταση ε, επιτακτική ε, πρέπει να ενθαρρύνουμε την ύπαρξη ορίων ταχυτήτων γιατί κάποιοι συνάδελφοι ε, διαφωνούν και το μπλοκάρουν αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω συνεχώς ότι υπάρχουν ε, ανθρώπινες ζωές που διακυβεύονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα ακόμη γεγονός ότι πάρα πολλοί ε, πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς. Υπάρχει, υπάρχουν προδιαγραφές για την κοινωνική ευθύνη των μέσων μεταφοράς, γιατί πρέπει πραγματικά αυτό το χάσμα μεταξύ των ε, απομακρυσμένων περιοχών και των ε, αστικών κέντρων να, μπορέσουν, να, να μπορέσει να γεφυρωθεί για να μην υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός. Πρέπει ε, τα μέσα μεταφοράς να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει αυτή την όθηση από κοινού με τις τοπικές αρχές για να μπορέσουμε να, να, να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ανάγκες των υποδομών τους και από οικονομικής απόψεως, στο πλαίσιο βέβαια της επικουρικότητας ε, ε, ενόψη της Συνόδου ε, για το κλίμα ε, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία ε, στην ενεργειακή αποδοτικότητα σε σχέση με την αστική κινητικότητα. Γι' αυτό εμεί προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο το δυνατόν συντομότερα να προτείνει ένα πακέτο ε, μεταφορών ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένοι σαφείς στόχοι για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίων. Κάποιοι συνάδελφοι εξακολουθούν ε, να ε, θεωρούν ότι δεν είναι πήγον αυτό ενώ είναι πήγον. Ζητούμε μείωση των κινητήρων, της χρήσης των κινητήρων από το 2030, των κινητήρων βενζίνης και δίζελ από το 2030 και ε, πλήρους κατάργησης μέχρι το 2050 Υπάρχει και το θέμα της χρήση των ορυκτών ε, καυσίμων στι αστικέ μεταφορές. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αντιμετωπίσει ε, πρέπει βασική προτεραιότητα να αποτελέσουν ε, σχέδια κινητικότητας βιώσιμα, αστικής κινητικότητας βιώ, βιώσιμα, τραμ, τελεφερίκ, ε, συνεπιβατισμός, ποδήλατο, όλα αυτά πρέπει να, να συνδυαστούν με τη διατροπικότητα. σας, στρέφομαι σε εσά κύριε Πρόεδρε, πρέπει να φροντίσουμε για το διπλασιασμό της χρήσης ε, του ποδηλάτου στις πόλεις μέχρι το 2025, όπως επίσης και την ενίσχυση των μέσων μεταφοράς με ορίζοντα το 2030. Γιατί δεν είναι μύθος ότι μπορεί κανείς να κάνει ποδήλατο στην πόλη. Γίνεται στην Κοπενχάγη. 55% ε, των ποδηλάτων ε, είναι στα αστικά κέντρα. Όλα αυτά μας δίνουν παράδειγμα και μας δίνουν κίνητρο για να ε, προχωρήσουμε. Βέβαια, σε τοπικό επίπεδο δεν υπάρχουν προγράμματα ε, βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ε, πρέπει να ε, βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης πρέπει να ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές να ε, θέσουν στο επίκεντρο τους πολίτες ε, των πόλεων ε, μέσω κατά το σχεδιασμό αυτών των αστικών κέντρων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, της συγχωρήπανσης, αλλά και το θέμα της μείωσης των ατυχημάτων. Υπάρχει βέβαια και το θέμα των μεταφορών, των αγαθών και εμπορευμάτων. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα και οπότε πρέπει να υπάρχει μια νέα αστική επιμελητία πράσινη, κάτι που είναι ε, βασικό, είναι ουσιαστική σημασία, κάτι το οποίο μας βρίσκει σε γενικές γραμμές αρκετά σύμφωνους. Ε, γιατί η βιώσιμη αστική κινητικότητα χρειάζεται επενδύσεις στις δημόσιες μεταφορές υπηρεσίες κοινή ωφελία. Ε, όταν η υποδομή είναι πάρα πολύ ακριβή πρέπει τουλάχιστον ένα τμήμα των εσόδων, για παράδειγμα της Ευρωβινιέτας ή των διοδίων να ε, χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας. Ζητώ λοιπόν ένα τμήμα των ε, ε, ταμείων, ζητώ από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, είτε του Ταμείου της Περιφερειακής Ανάπτυξης, είτε άλλων ταμείων να χορηγηθούν προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε το θέμα αυτής της αστικής κινητικότητας. Πρέπει να υπάρξει μια δυναμική στο πλαίσιο όλων των ε, σχετικών ταμείων. Και ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ξέρω ότι μερικές φορές έχουμε πραγματικές συζητήσει πολύ μακροχρόνιες κατά τη διάρκεια των ε, συμβιβαστικών αυτών τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πάντως και ελπίζω ολόκαρδα ε, ότι δεν θα είναι μόνο μία ακόμα έκθεση, αλλά θα είναι πραγματικά το αποτύπωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και ένδειξη ενός πραγμα... μιας πραγματικής κοινοβουλευτικής γενναιότητας, γιατί υπάρχουν προσδοκίες, υπάρχουν ανάγκες που έχουν εκφραστεί από πλευράς πολιτών, γιατί η κινητικότητα είναι κάτι που το ζουν κάθε μέρα, αλλά και από τους φορείς ε, του τομέα που περιμένουν πάρα πολλά από μας σήμερα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Ε, χαίρομαι πολύ που ε, ήμουν υπεύθυνη για την έκθεση αυτή. Θα συνεχίσω Την επόμενο, τον επόμενο μήνα θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και τον Νοέμβριο στην Ολομέλεια για την έκθεσή μου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, ε, κύριε Βέρκουνεν έχει το λόγο. Yes, thank you, Chairman, and thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτριά μας και όλους τους και εισηγητές. Ε, ήδη έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με την εισηγήτρια όλη Σκιώδης και από ό,τι φαίνεται θα χρειαστούν και άλλες συνεδριάσεις πριν καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. About urban mobility. Πολύ σημαντική έκθεση αυτή για την αστική κινητικότητα. Ξέρουμε ότι η αστιφιλία είναι παγκόσμια τάση, άρα η μετακίνηση στις πόλεις είναι όλο και μεγαλύτερο ζήτημα. Ξέρουμε ότι περισσότεροι Ευρωπαίοι ζουν στις πόλεις ήδη και υπάρχουν ε, πολλές δυνατότητες για το πώς μπορούμε ε, να κάνουμε τις μετακινήσεις στις πόλεις πιο ε, γρήγορες, πιο αποτελεσματικές και πιο ασφαλείς. Εμείς θέλουμε να ε, πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία η χωροταξία, η χρήση γης και η πολεδομία για να ε, δημιουργηθούν σωστά δίκτυα με καλή και γρήγορη μετακίνηση, βεβαίως λαμβάνοντας πάντα υπόψη και περιβαλλοντικά θέματα. Αυτές οι λύσεις ε, πρέπει να βρίσκονται από το σχέδιο του σχεδιασμού, γιατί έτσι είναι αηφόρες, και ε, έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια των μεταφορών, με τη ροή των συγκοινωνιών και με ε, τα διάφορα μέσα μεταφοράς. Ταυτόχρονα θέλουμε να τονίσουμε το σημαντικό ρόλο του σχεδιασμού, ε, αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, όλα αυτά τα ζητήματα συγκοινωνιολογίας και πολεδομίας. Καμιά φορά μάλιστα είναι και αρμοδιότητα της περιφέρειας, ή και των πόλεων. Εγώ είμαι από τη Φιλανδία. Ε, αυτά είναι ζητήματα, η πολεοδομία κατεξοχήν αρμοδιότητα των πόλεων, των δήμων. Βεβαίως ε, θέλουν και συμβουλές, αλλά όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα και από πόλη σε πόλη. Έχει μεγάλη σημασία να ε, σκεφτόμαστε και να ε, διαφυλάσσουμε την επικορικότητα. Όταν μιλάμε πάντα για πολεοδομία και αστικό σχεδιασμό, να μην μπαίνουμε πάρα πολύ στα χωράφια των πολιτών point of view is to use ε, υπάρχει επίσης και το θέμα των ευφυών μεταφορών και όλων των ε, τεχνολογιών που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, ξέρουμε ότι με έξυπνες λύσεις μεταφορών θα είναι πιο ασφαλείς, πιο γρήγορες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον ή συγκοινωνίες. Επίσης θα κάνουμε και οικονομία χρημάτων, διότι όλα τα προβλήματα μετακίνησης και κινητικότητας δεν λύνονται με νέες υποδομές κάθε φορά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο και πιο σοφό τις υφιστάμενες υποδομές και υπάρχει μεγάλο πεδίο εδώ δόξης λαμπρό ε, για τις ευφυείς και έξυπνες τεχνολογίες που ήδη διατίθενται. Η δική μας πολιτική ομάδα έκανε τροπολογίες φυσικά και αρκετές για τον εξή λόγο. Και εγώ προσωπικά θεωρούσα ότι το σχέδιο έκθεσης, πώς να πω, ήταν κάπως ανεδαφικό καμιά φορά δεν ήταν πάντα πάρα πολύ ρεαλιστικό και έβαινε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. <laughs> Θέλουμε να μείνουμε πιο γενικόλογοι, γιατί εμείς είμαστε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να σεβασόμαστε πάντα την επικουρικότητα και το ρόλο των πόλεων και των κρατών μελών και των περιφερειών. Ε, εμείς στόχους μπορούμε να βάζουμε, όχι δεσμευτικού βέβαια, αλλά να δίνουμε μια κατεύθυνση, να δείχνουμε το δρόμο για όλα τα κράτη-μέλη και μέχρι εκεί έτσι, προς τα που θα πρέπει να στραφούμε, αλλά να τους αφήσουμε την ελευθερία και τα χέρια τους ε, ελεύθερα για να αποφασίσουν πώς θα το κάνουν. Η δική μας πολιτική ομάδα ε, προσβλέπει στη συνέχιση συνεργασίας με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις, θα κάνουμε καλές συμβαστικές προτάσεις, περιμένετε ε, και προσβλέπουμε σε αυτό και στην επόμενη συνεδρίαση Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε περισσότερο για συμβιβασμού, αλλά έχει μεγάλη σημασία πάντα να σεβόμαστε την επικουρικότητα και να θυμόμαστε ότι είναι αρμοδιότητες όλα αυτά των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει τώρα εμεί να χαράσουμε δρόμου ή τη πολιτική στάθμευση θα πρέπει να έχει κάθε πόλη. Δεν είναι δική μα δουλειά αυτό. Ούτε πρέπει να πάρουμε εμεί τέτοιε αποφάσει. Γενικά, νομίζω θα βρούμε καλούς συμβιβασμούς τελικά ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο η έκθεση αυτή βασίζεται στη δουλειά που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο συμφωνώντας ε, για την Λευκή Βίβλο για την αναθεώρηση του τουρισμού. Γιατί πάρα πολλοί τομείς ε, που αναφέρονται επικαλύπτονται και πολύ σωστά η αστική κινητικότητα είναι ένα κομμάτι της ευρύτερης κινητικότητας και τα θέματα που ανέφερε η συγκεκριμένη είναι καθοριστική σημασία. Μίλησε πάρα πολύ για τα θέματα υγεία για την κρίση όσον αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας τη πόλη μας. Εμείς συμφωνούμε με όλα αυτά τα θέματα και η έκθεση αυτή πρέπει να τα εξετάσει όλα αυτά λεπτομαρώς. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια των δρόμων. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου περίπου 11.000 θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί ε, διαπιστώνονται κάθε χρόνο στις πόλεις μας. Βεβαίως ε, το θέμα δεν είναι ότι μπορούμε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε ε, καθαρά εθελοντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα ε, όριο ταχύτητας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πολλές φορές ε, είναι δυσάρεστο το ότι ξεπερνιέται αυτό το όριο ταχύτητας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Η συγγήτρια λοιπόν και η συνάδελφος επίσης από το ΕΛΚΑ ανέφερε και τα θέματα νομίζω της πολεοδομίας και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ε, η επικουρικότητα σίγουρα είναι κάτι που μας απασχολεί. Εμείς αυτό το εξετάζουμε στην Λευκή Βίβλο και είναι απολύτως ε, σαφές ότι η επικουρικότητα είναι σημαντική από την άλλη όμως υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που μπορούν να μα απασχολήσουν. χάρη, στην ε, Λευκή Βίβλο, ε, στην έκθεση για τη Λευκή Βίβλο, εκεί γίνεται λόγος ε, για το πώς η διαφάνεια θα πρέπει να είναι πιο συστηματική, κυρίως για πόλεις που έχουν ολοκληρωμένα συστήματα της πολεδομίας. Η επικουρικότητα δεν θα πρέπει να αναχαιτίζει το να γίνονται σωστά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες ακριβώς όπως το κάναμε και σε σχέση με τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές. Εξάλλου η δική μου η ομάδα υπογραμμίζει στις τροπολογίες τα δικαιώματα των εργαζομένων, το ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, μια πολιτική συμπερίληψης και όχι αποκλεισμού στις πόλεις. Ε, θέλουμε να πιστεύουμε το τελικό αποτέλεσμα θα παρουσιάσει τις θέσεις μας. Οι έρευνες που έχουμε κάνει εμείς σε αρκετές πόλεις, πρόσφατα στη Στοκχόλμη, έφτιαξαν τα θέματα που έχουν και με την κοστολόγηση των δρόμων για τη τελική ανάλυση το θέμα δεν είναι να ε, μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε αν δεν θίξουμε και κάποια σημαντικά πολιτικά θέματα. Η Τζόκι Φώστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τοζινόφσκι, ο σκιώδης μας δεν μπορούσε να ήταν εδώ, αλλά μου άφησε ένα σημείωμα για να κάνω ορισμένα ε, σχόλια εκ μέρους του θεωρεί ότι είναι μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση, είναι αυτή που πρέπει να έχουμε κατά τη σύνταξη αυτή τη έκθεση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το λέει αυτό γιατί είναι πρώην δήμαρχο πόλεο, οπότε προφανώ ε, έχει πείρα τοπική αυτοδιοίκηση, όπω πολλά μέλη τη Επιτροπή μα, ε, και μπορεί να δει ε, τι είναι πιθανό και τι δεν είναι τι είναι εφικτό και τι δεν είναι και μας υπενθυμίζει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία πολύ περιοριστικά ακριβώς επειδή υπάρχει η αρχή της επικουρικότητας και δεν μπορούμε να έχουμε μία λύση που να ισχύει για όλους, γιατί είναι πολύ διαφορετικές οι τοπικές συνθήκες και είναι κάτι το οποίο θεωρεί ότι είναι πρωταρχική σημασίας. Για αυτό το λόγο λοιπόν δεν ε, πιστεύει ότι μπορούμε να μπούμε ε, σε συζητήσεις ε, για τις αποφάσεις ε, σε επίπεδο κρατών μελών σε σχέση με τη διαχείριση των εσόδων από τα οδικά δίκτυα, από τις οδικές υποδομές ή για τα θέματα των ορυκτών καυσίμων. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν τι θα κάνουν με τέτοιου είδους έσοδα. Και τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία του σεβασμού της τεχνολογίας και της ουδετεραιότητας όταν πρόκειται για τα εναλλακτικά καύσιμα. Παρόλα αυτά, θα ήθελε να ευχαριστήσει την εισηγήτρια την κυρία Ντέλη για ε, την ε, εργασία της, ε, όπως επίσης και για τις συμβιβαστικές τροπολογίες και αναμένει αγωνίως την συζήτηση μαζί της. Ο κύριος Ματέης Φαν Μίτλβερκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και από πλευρά Σάλτε θα ήθελα να τονίσω και στα Ολλανδικά για αλλαγή θα μιλήσω πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και πόσο πρέπει να συζητάμε για μια βιώσιμη αστική κινητικότητα. Το είπαν όμως και άλλοι συνάδελφοι ε, εδώ πέρα είμαστε σε πολύ αλυσιρό έδαφος και είναι σαν να ε, κάνεις πατινάζ σε μια λίμνη που είναι πολύ λεπτό το στρώμα του πάγου. και Κινδυνεύουμε να πέσουμε μέσα στο παγωμένο νερό. Δεν θα πρέπει να υπαγορεύουμε πάρα πολύ στις πόλεις γιατί πρέπει να κάνουν δική τους αρμοδιότητα η αστική κινητικότητα. Οι δήμοι είναι δίπλα στον πολίτη. Εκείνοι ξέρουν. Δεν περιμένουμε να τους στείλουμε μαθήματα από τις Βρυξέλλες. Ε, ξέρουν πολύ καλύτερα τι πρέπει να κάνουν στις πόλεις οι ίδιοι. Αυτό που χρειάζεται είναι υποστήριξη από την Ευρώπη, όχι μαθήματα, υποστήριξη για το πώς μπορούν να χαράξουν μια στρατηγική και ένα σχεδιασμό χωρίς δεσμευτικές ε, ε, υπαγορεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταλλαγή ας πούμε γνώσης και πληροφοριών. Πώς μπορούμε τώρα στις πόλεις να έχουμε νέες μορφές κινητικότητας για να καταπολεμούμε ας πούμε τα μποτιλιαρίσματα και τη συμφόρηση. Για να είναι πιο καλή η συγκοινωνία και η μεταφορά, να μην υπάρχει υπερβολικό θόρυβο, να μην υπάρχουν υπερβολικέ εκπομπέ καυσαερίων, τέτοια πράγματα. Ε, αλλά ε, θα πρέπει να είναι στη διακριτική του ευκαιρία. Έτσι βλέπω εγώ αυτή την έκθεση. Υποστηρικτική προ του δήμου και τι κοινότητε, Θα πρέπει να δούμε τι συμβαστικέ προτάσει, όπω είπαν και οι προλαλήσαντε, να αποφύγουμε τι πάρα πολλέ ε, υποχρεωτικέ δεσμεύσει θα πρέπει εμείς να εστιάσουμε στις ευκαιρίες που έχουν οι πόλεις και λιγότερο στις υποχρεώσεις που έτσι και αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε, επαναλαμβάνω. Και χαίρομαι που το συζητάμε σήμερα, γιατί αυτή τη βδομάδα ξέρετε ότι είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο να συζητάμε και αυτά τα θέματα, να ανταλλάσσουμε απόψεις και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε ανθρώπους να είναι ποδηλάτε και αλλού στην Ευρώπη όπω και στι κάτω χώρε, Ξέρω ότι ο πρόεδρο είναι ένθερμος υποστηρικτή του ποδηλάτου, αλλά το θέμα είναι τι μπορούμε να πούμε και τι μπορούμε να προτείνουμε και τι να επιβάλλουμε. Εγώ το βλέπω ω κίνητρα όλα αυτά ε, και ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες να ολοκληρωθούν οι συμβιβαστικέ, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλέ τροπολογίε, το είπε και η συγκήτρια, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλέ ε, συμβιβαστικέ. 50 ε, παρακαλώ ε, στο στάδιο της προετοιμασίας. Και ξέρετε από τις 50 μόλις τις 13 έχουμε διεκπαιρεώσει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Αυτό που θέλουμε εμείς να στείλουμε ένα μήνυμα στις πόλεις και τίποτα να μην τους επιβάλλουμε. Αυτά και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η κυρία Μερία Κίλωνεν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης την εισηγήτρια και τους ε, σκέδους για την πάρα πολύ καλή συνεργασία. Η αστική κινητικότητα δεν πρέπει να υπερβάλλεται γιατί στην Ευρώπη ε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν στις πόλεις και η αισθηφιλία μοιάζει να είναι μελλοντική τάση. Εξάλλου η αστική βιωσιμότητα ευθύνεται για ένα μεγάλο κομμάτι των εκπομπών και των ε, ε, ατυχημάτων. Από την αστική κινητικότητα προκύπτουν και τα αιρούμενα σωματίδια τα οποία είναι υπεύθυνα για πάρα πολλές ε, βλάβες. Με τη συνάδελφο Ντέλη συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και με τους και και θα ήθελα στις δικές μου τις ε, τροπολογίες να προβάλλω τρία βασικά θέματα. Γιατί τώρα το 2015 μιλάμε πλέον για την αισθητική κινητικότητα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των πόρων. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση σημαίνει ότι δεν μπορούμε αυτά τα συστήματα να τα χρηματοδοτούμε περισσότερο. Ε, θα πρέπει να κάνουμε ακριβή χρήση, να κάνουμε σαφείς υπολογισμούς των κονδυλίων. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερα κονδύλια και να καταφεύγουμε στους ε, υπάρχοντες πόρους. Αυτό που έχει πει σημασία είναι ότι Η χρήση των ε, ιδιωτικών αυτοκινήτων των ΙΟΤΑΧΗ θα μειωνόταν, θα υπήρχε μεγαλύτερο ελεύθερο, περισσότερος ελεύθερος χώρος και μείωση των εκπομπών. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που βεβαίως ε, δεν έχει σχέση με τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εξευρεθούν νέες λύσεις για την ενέργεια. Η πράσινη ενέργεια μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στις αστικές συγκοινωνίες. Όταν αγοράζουμε νέα αυτοκίνητα και ίσως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι τα νέα καύσιμα και τα δίκτυα για νέα καύσιμα θα πρέπει να τα εντάσσουμε μέσα στην υποδομή των μεταφορών. Στην Επιτροπή μας θα πρέπει να ακούμε περισσότερο και τους χρήστες, τη δική τους τη φωνή, και να μην ξεχνάμε να έχουμε κατά νου ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά διότι για αυτά τα νέα ε, πρότυπα υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια χρήστες ε, στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου, γιατί αλλιώς υποτιμούμε τους χρήστες και τους πολίτες. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι οι ευφυείς αστικές ε, συγκοινωνίες δεν έχουν σχέση μόνο με τις μεγάλες πόλεις, αλλά με τις ε, μικρομεσαίες. Ο κύριος Πέτερ να έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρέπει να δούμε πάρα πολύ τι γίνεται με την αστική κινητικότητα. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα συμφόρησης και 30% ε, των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ε, συμβαίνουν στις πόλεις. Θα πρέπει να το καταλάβουμε. Βλέπουμε πως έχει κατάσταση και εδώ στο Βέλγιο που ζούμε. Δεν ξέρω, κοιτά, έχετε δει πως οδηγούν εδώ οι άνθρωποι. Νομίζουν ότι έχουν κληρονομήσει το DNA του Μίχαλ Σούμαχερ. και ε, ούτε άμα κορνάρεις θα φύγουν τα ποτηλιαρίσματα. Ε, δεν ξέρω, έχω μεγάλο πρόβλημα με τη συμφόρηση την κυκλοφορία εκεί στο Βέλιο. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουν τα συστήματα για να μπορούμε ε, ίσως τα εμπορεύματα ας πούμε να τα παραδίδουμε τη νύχτα για να μην έχουμε περισσότερη επιβάρυνση και συμφόρηση στις πόλεις από φορτηγά που ή φορτηγά που κυκλοφορούν στις πόλεις τη μέρα για να μοιράζουν τα εμπορεύματα. Δεν ξέρω, στη Φιλανδία και στη Σουηδία χρησιμοποιούνται ίδια άλλα συστήματα. Χρειάζονται φορτηγά για να διανέμεις ένα εμπόρευμα από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β στην πόλη. Δεν πας από τη βόρεια στη νότια Γερμανία σε ένα αυτοκινητόδρομο για να χρειάζεσαι φορτηγό. Μέσα στην πόλη χρειάζεσαι ολόκληρο φορτηγό τέτοιου μεγέθου για να μεταφέρει εμπορεύματα. Αυτά όλα θα πρέπει να τα ξέρουν τα κράτη-μέλη, να ε, έχουμε προτάσει, όχι εναρμόνιση φυσικά, αλλά για να μπορεί ο καθένα να καθορίζει την πορεία του και να ε, χρησιμοποιεί αυτό που τον εξυπηρετεί και τον βολεύει. Πολλά είναι τα θέματα και τα ζητήματα, αλλά Συμφωνώ απολύτως. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Τώρα λοιπόν ολοκληρώθηκε ο γύρος των σχεδόν εισηγητών. Είμαστε λίγο υπό πίεση χρόνου γιατί η Επίτροπος θα έρθει στις 5 και 20 και έχουμε άλλο ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Ένα λεπτό παρακαλώ. Η κυρία Κριστίν Ρεβονταλών, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Καριμά και τους κοιόδης ηγητές για την έκθεση αυτή. Είναι πραγματικά αποφασιστική σημασία και χαίρομαι που οι συζητήσει είναι πάρα πολύ εντατικέ και θέλουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας τον Οκτώβριο και στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο για να προλάβουμε τη διάσκεψη COP21 γιατί θα ήταν κρίμα να μην έχει ψηφιστεί αυτή η έκθεση πριν την COP21. Ξέρουμε ότι οι αστικές συγκοινωνίες οφείλονται κατά 21% για την κλιματική αλλαγή και έχουμε ε, μια τεράστια πρόκληση ενώπιον μας. Αυτή η κινητικότητα να γίνει υποδειγματική ε, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Έχει λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω για αυτά που λέτε για την επικουρικότητα, αλλά δεν θα πρέπει να είναι αυτό ένα εργαλείο για να μπλοκάρουμε τη συζήτηση στην Ευρώπη για την αηφόρο κινητικότητα. Κανείς δεν αμφισβητεί ε, την περιφερειακή ή την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ είμαι περιφερειακή σύμβουλος στην Ile de France και είμαι και σε ένα συμβούλιο μεταφορών επίσης μέλος στη Γαλλία. Τα ξέρω όλα αυτά. Ε, ξέρω ε, ότι χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ένα πλαίσιο για να πάρουν τις αποφάσεις οι αρμόδιοι Οπωσδήποτε ε, ε, υπάρχουν και τα κοινωνικά ζητήματα εδώ για να ε, σταματήσει αυτό το ρήγμα, το χάσμα μεταξύ των διαφόρων περιοχών αστικών ή μη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να είμαι αυστηρό γιατί δεν θα προλάβουμε αλλιώ. Ο Γιάννη Νίλσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος συμμετέχει στη συζήτηση αυτή. Γιατί? γιατί σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις πόλεις έχουμε ένα πρόβλημα με τους, για τους πολίτες, είναι κάτι που τους ενδιαφέρει. Ε, όλους όσους ε, εργάζονται σε τοπικό επίπεδο, εγώ και 15 χρόνια μιλάω για τις βιώσιμες πόλεις, πώς είναι δυνατόν να τις καταστήσουμε βιώσιμες τις πόλεις. Χρειαζόμαστε καθοδήγηση, χρειαζόμαστε ανταλλαγή εμπειριών. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών μας έδωσε κίνητρο και αυτό έγινε με την εβδομάδα της κινητικότητας που προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Πολλές πόλεις αντάλλαξαν τις εμπειρίες τους. Υπάρχει και ε, διαγωνισμός αυτή τη στιγμή ε, επιλογής της πόλης που τα καταφέρνει καλύτερα από απόψεως αστικής κινητικότητας. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι, θα έλεγα ότι το Έστασουντ είναι η καλύτερη πόλη. Ευχαριστώ που τηρείτε και το χρόνο. Ο κύριος Κόχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα να ευχαριστήσω την Καριμάντελη για τη δουλειά της που ήταν και πάρα πολύ και προσβλέπω στη μεγάλη της προθυμία για συμβιβασμούς. Το θέμα είναι βιώσιμη αστική ε, κινητικότητα όχι των μεγάλων αστικών κέντρων. Προσοχή, δεν μιλάμε για μητροπολιτικά κέντρα. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας και αυτοδιοικητικός και ε, μου είναι ιδιαίτερα προσφυλής η επικορικότητα και όταν στο σημείο 3 μιλάμε για ιεράρχηση των ε, συγκοινωνιών στο 18 τα εμπορικά κέντρα κτλ θέλουμε να τα ρυθμίσουμε που θα εδρεύουν ή να έχει κατευθυντήριες γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χώρους στάθμευσης και τα λοιπά και χρήση στο κέντρο, αυτό νομίζω ε, είναι κάτι υπερβολικό. Ούτε είναι δική μας δουλειά να πούμε αν θα είναι δωρεάν οι συγκοινωνίες οι αστικές και τα ΕΦΗ e συστήματα και ε, το ενιαίο εισιτήριο και η τιμολόγηση μου λείπει και έχω κάνει προτάσεις αντίστοιχες που ελπίζω να ληφθούν υπόψη και να μπορέσουν να ενταχθούν στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και για την τήρηση του χρόνου. Το λόγο έχει ο Βιμ Φαντεκάμπ. Οι δύο προηγούμενοι τήρησαν το χρόνο. Πρόσεχε. Πρόεδρε, γνωρίζετε πόσο λακωνικός είμαι πάντα. Το κείμενο, ε, το, το θέμα μάλλον το έχω παρακολουθήσει εδώ και ένα χρόνο τώρα και φοβούμαι ότι η συγγήτρια εκτοξεύει πολλές απειλές και, ε, και μιλάει λίγο για ευκαιρίες. Η βιώσιμη αστική κινητικότητα έχει να κάνει και με την καινοτομία και με την οικονομία και με την επικουρικότητα. Δεν είναι μόνο απειλές. Και θα ήθελα αυτά τα στοιχεία λίγο να τα δω να τονίζονται περισσότερο στην έκθεση. Αυτά ε, τα είπε και ο συνάδελφος από τους φιλελευθέρους. Όταν γίνεται λόγος για τη ρήπανση, για τη δημόσια υγεία και για την ασφάλεια, αυτά είναι τα σωστά θέματα. Αλλά ηλεκτρονικές συγκοινωνίες στην πόλη. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα με το ποδήλατο. Αυτό είναι λάθος ρομαντισμός. Ε, θέλω μεγαλύτερη προσοχή λοιπόν για τις ευκαιρίες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια για τις πόλεις ε, και ε, να, λίγη περισσότερη προσοχή για την οικονομία και σας χαρίζω και δύο δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ θαυμάσια. Ε, γιατί όλα ε, τα καλά πράγματα είναι τρία, οι τρεις ομιλητές τα τήρησαν και τώρα η κυρία για άλλα. Θα προσπαθήσω. Ε, συγχαρητήρια στην κυρία Ντελή ε, για, για τους συμβασμούς. Από τη μια κατανοώ αυτό που μιλάει ε, για αστικά διόδια, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και ποια είναι και η κοινωνική δομή σε ορισμένες χώρες και στη δική της. Ε, κανονικά οι νέοι που έχουν λίγα λεφτά και οικογένειες, η εργατική τάξη έχει εξοφηθεί ε, εκτός των πόλεων και τώρα τους ζητάνε αστικά διόδια για να μπουν στην πόλη. Αυτό με τα ποδήλατα είναι ωραίο και καλό, αλλά θα πρέπει να συμφιλειωθεί με τους πεζούς. Σε ορισμένες πόλεις δεν είναι τόσο εύκολο ε, και για τους εργαζόμενους. Μιλάει η ίδια για μια ειδική επιτροπή. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ενισχυθεί η Γενική Επιτροπή Διαλόγου ε, για ε, τις μεταφορές. Τα κονδύλια δεν τα ανακαλύψαμε σήμερα για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη στο σχέδιο Juncker. Ήδη στα διευρωπαϊκά δίκτυα υπήρχαν και ε, τα αστικά κονδύλια και τα αστικά προγράμματα μπορούν να μπουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα και μπήκανε, ακόμα και αν δεν ήταν της αρισκίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δομινίκ Ρικέ. Πολύ σύντομα. Καταρχάς, ε, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε με τις διαπιστώσεις ε, και τις ανησυχίες ε, της συζητήτριας. Κάνει μία μακροπρόχρια πρόβλεψη που είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όμως, υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ των αστικών κέντρων και των διαφόρων προβλημάτων για λόγους πολιτικών, για το κλίμα των κρατών μελών και Επίσης, οι αλλαγές που ε, διαπιστώνουμε προκύπτουν από την ίδια την κοινωνία και από την επιστημονική πρόοδο. Οπότε όλα αυτά τα πολύ περιοριστικά που αναφέρεται μπορεί να ε, ε, ισχύει ε, στο, για, στην δική της, ε, για τη δική της θεώρηση όμως υπάρχουν και τα μοντέλα τα οποία μόλις αναφέρθηκαν γιατί άλλαξε η οργάνωση της, κοινων, της κοινωνίας και γι' αυτό πιστεύω ότι ε, το, η έκθεση είναι εκτός τόπου και χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνεται η ανάλυση ε, για την αστική κινητικότητα, το θέμα του κλίματος. Πολύ ωραία περιγράφονται όλα αυτά και εκεί μάλιστα όπου αναφέρεται ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα, να παρουσιάσουμε τις βέλτιστες ε, πρακτικές, να ασχοληθούμε με ευφυείς ε, τεχνολογίες, όλα αυτά είναι πολύ καλά, τέτοιου του σχέδια μπορεί κανείς να τα ανταλλάξει. Όσον αφορά όμως τις αρμοδιότητες και τα ρυθμιστικά, εκεί υπάρχει κάποιο λάθος. Εμείς είμαστε που βάζουμε το πλαίσιο, ε, βάζουμε στόχους για το διοξείδιο του άνθρακα και πρέπει μετά αυτοί οι στόχοι να, ε, να εφαρμοστούν. Όμως εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε και δεν παρεμβαίνουμε στις αρμοδιότητες ε, τις εθνικές και τις ε, περιφερειακές. Ε, είχαμε εκλογές στη Βόρεια Βεσφαλία και σας λέω ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα τα αντιμετώπισαν εκείνοι που δεν είχαν οργανώσει σωστά τις αστικές τους συγκοινωνίες. Δηλαδή η πολιτική και η οικονομική ευθύνη για την οργάνωση του προσωπικού των αστικών συγκοινωνιών είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά και μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε όσον αφορά το όριο ταχύτητα ή τον προγραμματισμό. Αυτό δεν επιτρέπεται ούτε και σαν συμβιβασμό. Η κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ πολύ να συνεχίσω. Λέξαν πάρα πολλά για την επικουρικότητα. Πράγματι, πολύ σωστά θα πρέπει να προβούμε σε βελτιώσεις. Εγώ, ας πούμε, πιστεύω ότι αυτό το EPNV θα ισχύει μέχρι το 30. Τέλο πάντων, εγώ θεωρώ γενικότερα ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Το να επιβληθεί παντού η ταχύτητα 30 χιλιόμετρων, δεν ξέρω αν αυτό είναι η λύση ή αν είναι καλύτερα να υπάρχουν ευφυή συστήματα. Αυτό είναι πιο έξυπνο και υπόθηκε προηγουμένως και από συνάδελφο, θα πρέπει να ακούμε και την άποψη του χρήστη, του καταναλωτή, του επιχειρηματία, που και αυτοί υποτίθεται θα εξοπλίζουν τις πόλεις. Δεν γίνεται να γίνεται η κυκλοφορία μόνο με ποδήλατα, χρειαζόμαστε στις πόλεις και μικρά φορτηγά. Και αυτό θα πρέπει να είναι εφικτό, να αναζητήσουμε κάποιες καλές λύσεις. Αλλά, εν περιπτώσει, Λοιπόν, κοιτάξτε, το 70% όλων των εκπομπών που είναι διοξείδιο του άνθρακα προέρχονται από τις μεταφορές, από την κυκλοφορία. Εκεί υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία και υπάρχουν αναλύσεις. Ας πούμε στο Βερολίνο σε 10 χρόνια διπλασιάσαμε τα ποδήλατα. Πολλοί δεν έχουν πια αυτοκίνητο και το 50% ε, των ε, εμπορευματικών μεταφορών θα μπορούσε να μεταφέρεται με e-bikes, ηλεκτρονικά ποδήλατα. Το θέμα είναι πώς θα τα προάγουμε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πει τα χρήματα να επενδυθούν στο ε, σωστό επίπεδο και όχι στο λάθος. Για το ταχύτητα 30, κύριε Πίπερ, την προηγούμενη θητεία αποφασίσαμε αυτό να είναι η τακτική κανονική ταχύτητα και οι πόλεις να αποφασίσουν μόνοι τους που θα μπορεί το όριο να είναι υψηλότερο. Ε, αυτό το δέχτηκαν όλοι οι ε,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 Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερη. Καταρχά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι σε αυτό το σημαντικό θέμα στην Επιτροπή σα. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, αλλά όλου εσά που καταθέσατε τι 502 τροπολογίε. Πραγματικά είναι ένα πολύ εντυπωσιακό αριθμό και ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε 50 συμβιβαστικέ τροπολογίε που θα τύχουν τη υποστήριξη όχι μόνο αυτή τη Επιτροπή, ε, αλλά ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί Όλο αυτό το ενδιαφέρον και ε, όλα αυτά τα σχόλια θεωρώ, θα τα θεωρώ ε, ως ε, απόδειξη της σημασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της αστικής κινητικότητας, βιώσιμη αστικής κινητικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και για μας αλλά και για τις τοπικές και περιφερειακές ε, αρχές. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί έχετε ξανακούσει τις απόψεις μου για το θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, Καλό είναι να ακούμε ότι συμφωνούμε στο ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα ε, τα οποία πρέπει να μας αποσχολήσουν στο πλαίσιο της αστικής κινητικότητας. Δεν είναι μόνο η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αντίκτυπο στην υγεία, κλιματική αλλαγή ε, όσων ζουν στις πόλεις, αλλά η σημασία των πόλεων ε, ως στοιχείων ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να είμαστε επιτυχείς πρέπει να έχουμε επιτυχημένες πόλεις. Γι' αυτό ακριβώς ακούσατε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναφέρεται συγκεκριμένα στις πόλεις, να απευθύνεται στις πόλεις ε, και νομίζω ότι είναι ένας από τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ε, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Όμως οι πόλεις ε, έχουν να κάνουν και με την ανάπτυξη και με τις θέσεις απασχόλησης. Πρέπει να είναι μια ε, θετική λύση που όταν μια θετική λύση εφαρμόζεται σε μια πόλη μπορεί να δοκιμαστεί και σε μια άλλη πόλη. Μας, ε, είμαστε ιδιαίτερη ευαίσθητοι για το θέμα της επικουρικότητας. Δεν είναι ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των εθνικών κυβερνήσεων να πούν σε κάθε μία από τις πόλεις πώς πρέπει ε, ποια προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουν και ποια πρέπει να επιλύσουν. Ε, ο, ο ρόλος μας είναι να έχουμε μέσα και εργαλεία και να τους πούμε πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό ακριβώς η ανταλλαγή καλών πρακτικών και καλών ε, ιδεών, ιδεών ενίσχυση της ανάπτυξης των προγραμμάτων των, της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, χωρίς τους υποχρεώνουμε να τα εφαρμόσουν, είναι εργαλεία τα οποία μα δίνουν τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια περιεκτική και καλά οργανωμένη, σε ένα περιεκτικό και καλά οργανωμένο σχεδιασμό για το μέλλον, όπω για παράδειγμα ε, προγράμματα το 2020, ε, το συνδέοντα στην Ευρώπη, η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, όλα αυτά πρέπει να είναι σωστά στοχευμένα, ώστε να βοηθήσουμε τις πόλεις να επιτύχουν αυτού του στόχου που έχουμε συμφωνήσει. Να σα ευχαριστήσω που πολλέ φορέ αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ε, Παράγματι ε, θα γίνει έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έναρξή της, τα εγγένειά της και θα είναι μία ακόμη ευκαιρία να πούμε στις ευρωπαϊκές πόλεις και στους πολίτες ότι υπάρχουν ήδη λύσεις Μόνο πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουν την υποστήριξη και τα μέσα να εφαρμόσουν τις λύσεις σε αυτές τις πόλεις τους, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται αυτές οι πόλεις, ε, ποια είναι η γεωγραφία τους, ποια είναι η οικονομική τους κατάσταση και ποιο είναι το μέγεθός τους. Θα ολοκληρώσω γιατί δεν θέλω η Επιτροπός μας ε, να ε, περιμένει, όπως δεν θέλετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα σχόλια. Η κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, για όλες αυτές τις παρατηρήσεις, οι οποίες όμως χρήζουν απαντήσεων. Καταρχάς, όλοι συμφωνούμε για τις ευφυείς μεταφορές, ε, αναφέρθηκε το θέμα του συνεπιβατισμού, αλλά η ευφυείς μετακίνηση, και επανέρχομαι σε αυτό που είπε το ΕΛΚ, μία αστική μεταφορά δεν γίνεται εάν δεν βελτιστοποιήσουμε το θέμα των υποδομών, των μεταφορών, ε, τη χρήση του χώρου κλπ. κλπ. Όλα αυτά τα θέματα θέματα ε, του άθεος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αφορούν την κινητικότητα του αύριο. Και επανέρχομαι στην παρατήρηση του Ντομινίκ Ρικέ, γιατί μας είπε, μα ε, δεν είναι δυνατόν, είναι εκτός τόπου και χρόνου η έκθεση. Όχι, έχουμε μια διαπίστωση μέσα αυτής της έκθεσης και λέμε πώς είναι δυνατόν εφιώς να δημιουργήσουμε την πόλη του αύριο. Με, με με τους πόρου που έχουμε. Όμως κάποια στιγμή πρέπει να πάμε παραπέρα. Και όταν μου λέτε, και εδώ διαφωνώ, ότι ναι, μα έχουμε την επικουρικότητα, μα εγώ δεν είπα την έκθεσή μου ότι πρέπει να πάμε πέρα από τις πόλεις και πέρα από τα κράτη. Ενθαρρύνει, ενθαρρύνει απλώς και ποια είναι η, άποψη των χρηστών μας λέτε. Μα οι χρήστες είναι αυτοί που λένε ότι θέλουμε 30 χιλιόμετρα την ώρα γιατί το θέλουμε, γιατί διακινδυνεύουμε τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας. Μην μου λέτε λοιπόν σήμερα ότι δεν υπάρχει σύνδεση με τους χρήστες. Όχι, αυτό δεν ισχύει, αυτό ακριβώς προσπαθώ να επιτύχω. Δεύτερο θέμα που είναι σημαντικό για μένα, βεβαίως ανταλλαγή εμπειριών κλπ. Είναι μία από, από τα βασικά καλά στοιχεία αυτής της ε, έκθεσης. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Και ένα τελευταίο ε, σημείο για την κινητικότητα. Σήμερα προχωρά με, μια, με ένα τεχνολογικό ρυθμό πάρα πολύ γρήγορο, ε, μιλάμε για το Google Car, μιλάμε για τόσα πράγματα. Ε, σε αυτό πρέπει να προσαρμοστούμε, γιατί πρέπει και ε, η αυτοκινητοβιομηχανία να προσαρμοστεί στον αυριανό κόσμο. Πρέπει να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα εν ώψη τη Συνόδου για το κλίμα, αλλά και στο πλαίσιο των ευθυνών που έχουμε στην Επιτροπή μας. Δεν θα κάνουμε κάθε χρόνο έκθεση για την αστική κοινότητα. Αλήθεια είναι αυτό που λέω για την αστική κινητικότητα. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε ένα βασικό πλαίσιο, να έχουμε ένα χάρτη πορείας που θα προτείνουμε στις πόλεις για να, μπορούν, να μπορούμε στο πλαίσιο της Ευρώπης να έχουμε ένα όραμα ε, μιας επιθυμητής πόλης και μιας βιώσιμης κυρίως πόλης, γιατί δεν θα είναι βιώσιμη πια οι πόλεις μας αν δεν κάνουμε τίποτε για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνεδρίαση και ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών που είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη ε, της Επιτροπής πλην όμως και κλεισμένων των θυρών. Έτσι, μόνο οι συντονιστές και τα μέλη της Επιτροπής αν επιθυμείτε, αλλά όχι το κοινό.